Meine Damen und Herren, ich darf... Ο πρόεδρος Μπροκ. Καλή σας μέρα. Κυρίσω την έναρξη της τελευταίας συνεδρίασης προ του Πάσχα. Θα ακούσατε σίγουρα ότι προ μια ώρα περίπου συνέβη απόπειρα, επίθεση στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Φαίνεται πως έγινε στο check-in της εταιρείας American Airlines. Ε, φαίνεται πως υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί. Αντιλαμβάνεστε, βλέπουμε όλοι δηλαδή ότι η τρομοκρατία πλώνει τα πλοκάμια της παντού και εκεί όπου εμείς οι ίδιοι δραστηριοποιούμεθα. Και σήμερα το πρωί που πέρασα από εδώ Υπάρχει πολύ ανοιχτός χώρος, ενώ ανάμεσα στα δύο κτίρια μπορεί να περάσει ολόκληρο φορτηγό αυτοκίνητο. αν το φορτηγό αυτοκίνητο μεταφέρει και μερικές βόμβες, δεν θα μείνει τίποτα από το κοινοβούλιο, έτσι. Αντιλαμβάνεστε, ανοιχτή πρόσβαση. Παρόλο που οφείλω να αναγνωρίσω ότι το κοινοβούλιο, η διοίκηση του κοινοβουλίου δηλαδή, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Αλλά αυτό το μέρο δεν είναι αρμοδιότητα του κοινοβουλίου, είναι των αρχών των Βρυξελών. Σας παρακαλώ να εγερθείτε για ενός λεπτού σιγή για τα θύματα αυτής της δημοκρατικής επιθέσεως. Herzlichen Dank, dass Sie sich erhoben haben. jetzt der Bericht. Με συγχωρείτε, ορίστε. Εγώ νομίζω ότι αποδίδεται τιμή στους τρομοκράτες διότι ταυτόχρονα τουλάχιστον 12 νεκροί υπάρχουν από τροχαία ατυχήματα. Δεν υπάρχει κανένας ειδικός λόγος να Αποδίδετε τιμή στους τρομοκράτες. Αυτό κάνετε. Ο πρώτος μπλοκ. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι οι παρατηρήσεις σας στρέφονται κατά των ίδιων των εαυτών τους. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην ημερησία διάταξη για την Αλβανία. Κύριε Φλέκενστάιν, έχετε καμία παρατήρηση ή τι έχετε εξαντλήσει πλέον όλες. Μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρίζω σελίδα. Τροπολογία 40, συγγνώμη, όχι 44, λέει ο πρόεδρος, κάτι άλλο. 40, τροπολογία 40. Υπέρ με προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πώς θα ψηφίσετε εσείς, ναι ή όχι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 28 υπέρ 27 κατά. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 με προφορική τροπολογία Φλέκενστάιν. Δεν έχει πει υπέρ ο πρόεδρος. Α, ο κύριος Φλέκενστάιν. Σε συμφωνία κύριε πρόεδρε με τον κύριο Κούκαν του Λαϊκού Κόμματος επιθυμούμε να αφαιρεθούν οι λέξεις and its enforcement. Γιατί δεν θέλουμε να προκληθεί ασφαλμένη εντύπωση ότι δηλαδή μόνο όταν πια θα έχουν εφαρμοστεί πλήρω όλε αυτέ οι μεταρρυθμίσει θα μπορούν να αρχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Αυτή, η ευθύνη το έτοιμά μα. Ευχαριστώ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Την 6 την ψηφίσαμε μόλις. Α, ο συμβαστική 6 λέει ο πρόεδρος τώρα. Υπέρ κατά αποχές. Μα την ψηφίσαμε όμως. Συμβαστική 7. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91, το πρωί 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζει 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98, 98 υπέρ. Κατά. όχι, Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κάποιος ζητεί επαλήθευση. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 31 κατά απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σύμβα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ακολουθεί η προφορική τροπολογία 3 ψηφί υπέρ κατά Επαλήθευση παρακαλώ. Πέραση της ψήφου. 36 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά γίνεται, ε, εγκρίνεται του κ. Πίτσουλα ενάντια στη ψήφου της ομάδας του. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. 163 επαναλαμβάνει προς 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται Check, επαλήθευση δηλαδή, ηλεκτρονική. 10, υπαριθμόν 10. Πέρας. Ψήφι 32 υπέρ, 23 κατά. Άρα σωστά είπα ότι υπερψηφίστηκε. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Πέρας της ψηφοφορίας. «48» μαζί με τον κύριο Μπιλαμόν υπέρ, 3 κατά 4 αποχές. Και ακολουθεί η έκθεση για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Κύριε Ισηγητά, έχετε κάτι να σημειώσετε. Όχι. Άλλωστε δεν με ακούτε. Ούτε καν με ακούτε. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στην συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι ε, απαιτεί τη ηλεκτρονική παλήθευση, αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Τέλος. 30 ψήφοι υπέρ και 25 κατά. Ορίστε. Ο κύριος Πρέντα επιθυμεί να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, μάθαμε ότι και στο μετρό μόλις έγινε μία έκρηξη. Όπως καταλαβαίνετε, με ιδιαίτερη θλίψη τα μαθαίνουμε όλα αυτά. Έκρηξη στο μετρό. Τέλος πάντων, θα τελειώσουμε την ψηφοφορία, αλλά όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση Also mein Vorschlag Ο πρόεδρος Πρόκ, η πρότασή μου είναι η εξή. Ήδη αγερθήκαμε για ενός λεπτού σιγή, αλλά δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να διακόψουμε τις εργασίες μας λόγω των τρομοκρατών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία και με την ημερησία μας διάταξη. Θα παρακαλέσω την γραμματεία να αναζητήσει κάποιον ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει πληρέστερα. Ίσως κάποιος από τις αρχές ασφαλείας να μας κάνει μια προσωρινή ενημέρωση για τα τεκτενόμενα. Συνεχίζουμε λοιπόν. 167 την ψηφίσαμε. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. 31 ψήφοι υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Επανάληψη. 65 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 πρώτο μέρος, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί η τροπολογία 109 πρώτο μέρος, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα επίσης. Μάλιστα, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση.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 αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά. Επαλήθευση, αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Σας παρακαλώ ωστόσο. Παρά την ψυχολογική επιβάρυνση να συμμετέχετε στην ψυχοφορία. και εγώ ο ίδιος προσωπικά ε, έχω δυσκολία να συγκεντρωθώ γιατί οι σκέψεις μου είναι αλλού. Αλλά αν ψηφίζετε όλοι θα μπορώ να διακρίνω καλύτερα τις πλειοψηφίες. Έληξε η ψηφοφορία 31 υπέρ 24 κατά. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το Λαϊκό Κόμμα δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. Λοιπόν, ξανά, 145 υπέρ. Επαναλαμβάνω. Κατά, λοιπόν. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές αυτό εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ Ω, με συγχωρείτε, πρώτα 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται 32 ψήφοι υπέρ 21 κατά. Πέτ 159 δηλαδή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμόν 5 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κύριε Καν. Ενίσταμε κατά της ε, προφορικής αυτής τροπολογίας, διότι δεν προσθέτει τίποτε, η δε διατύπωση είναι παρόμοια με αυτήν που ήδη έχουμε προτείνει εμείς. Άρα τότε θα ψηφίσουμε μόνο την 5 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ της 5. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μόλις ακούσαμε ότι έγινε και άλλη έκρηξη στο Σουμάν. Στο σταθμό του μετρό υποθέτω, υποθετή. έμεινες. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψήφι 27 υπέρ 26 κατά. Υπαριθμόν 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 και 2. Σε σπάνιο συντονισμό Μακάριστερ Πέτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου. Τέλος. Ο Πρόεδρος. Θα διακόψω την συνεδρίαση για πέντε λεπτά και παρακαλώ να προσέλθουν οι συντονιστές. Έγινε άλλη μια επίθεση μεταξύ Σούμαν και Μάλμπεκ. Απ' έξω έχουν κλείσει οι είσοδοι του Κοινοβουλίου τώρα. Και είμαστε σε επαφή με το Γενικό Γραμματέα για να δούμε τι θα κάνουμε. Προτείνω να διακόψουμε ακόμη για πέντε λεπτά για να έλθουμε σε επαφή με τα γραφεία μας να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Σε, σε, 5 λεπτά, σε 5 λεπτά θα αρχίσουμε την ψηφοφορία.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 Is that also by my Δεν λειτουργεί το κινητό μου. Δεν υπάρχει... Φαίνεται πως δεν υπάρχει δίκτυο πλέον. 62 δύο, Γκάλερ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόκειται για την έκθεση της κυρίας Καλνιέτε. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Πέρασε. ...26 ψήφοι υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, Επαλήθευση. Πέρασε. 24 υπέρ 28 κατά εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος αλλά έκανε λάθος προφανώς. Με συγχωρείτε όχι μου φάνηκε ήταν 23 λέει ο πρόεδρος. Αν είχα καλύτερα γυαλιά δεν θα μου συνέβαινε αυτό. Άρα απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι με συγχωρείτε, εγκρίνεται. 83 ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Δεν ψηφίζει η σοσιαλιστική ομάδα. Πέρας. Ψήφι υπέρ 33 κατά 17. Εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά. Όχι κύριε Πρόεδρε, 90. Α, την επαλήθη κάναμε στην 87. Λοιπόν, ωραία. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Τέλος. 18 υπέρ 33 κατά απολύτεται. Συμβαστική 5 κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 ναι. 142 ναι. σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. 142 όπως είπα έχει δύο τμήματα. Ένα και δύο. Το πρώτο λύγει με τις αγγλικές λέξεις Union Budget και το δεύτερο The EDA. Το πρώτο ενεκρίθη, το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Τέλος. <clears throat> Τέλος. Ψήφι 13 υπέρ, 38 κατά, απερίφθη. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά Μόλις 10% ε, των βουλευτών συμμετέχουν. 157 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές επαναλαμβάνεται 178 υπέρ κατά αποχές, α, δεν είπε αποχές ο πρόεδρος εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση Πέρας. Ψήφι 25 υπέρ 26 κατά απορρίπτεται. 188 υπέρ. Με συγχωρείτε, 183 υπέρ. Υπέρ λέω. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τέλος. Ψήφι 29 υπέρ 22 κατά. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εκατόν ενενήντα υπέρ. Θέλετε επαλήθευση για το 190. Θα επαναλάβουμε το 190 λοιπόν, δεν πειράζει. 26 ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Ενεκρίθη λοιπόν. 191 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ας, ας επαληθεύσουμε. Ας επαληθεύσουμε. Δεν είμαι σίγουρος. Απορρίπτεται εν τέλει. 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν όπως ε, σας είχα πει. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 247 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ας την επαληθεύσουμε καλύτερα. 2.47 πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. επαλήφθηση μάλιστα. Απερίφθη. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 267 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε 267 δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα τέλος με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω με, μικρό, με μικρή διαφορά αλλά ας την επαληθεύσουμε. 283 Τέλος. Απερίφθη. Αυτή τη φορά με μία ψήφο διαφορά. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχω δυστυχώς άλλη επιλογή, πρέπει να επαληθεύσουμε. Τέλος. Απερίφη 25-24. 292 υπέρ κατά αποχές. Σύντομη ηλεκτρονική παρήθευση πάλι. Είναι πολύ μοιρασμένο το σώμα. Πέρασε. απερίφθη. 293 και 94 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 295 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, ορισμένοι δεν σηκώνουν και το χέρι καλά και δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. ψήφο διαφορά. 200 διακόπτει κάποιος βουλευτής, αλλά δεν ακούμε τι λέει. Όχι, καλώς. Λοιπόν, <clears throat> είναι κρίση 295 παιδιών. 296 του κ. Πρέντα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 302 υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση. Επαλήθευση και πάλι. 302. 24 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Τέλος. Απερίφθη 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Θέλετε παρήθευση τώρα. Καλώς λοιπόν. 306 beauty coffer. Επαλήθευση. Απερίφθη. 307 και 308 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 310. Against abstentions adopted. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ κατά αποχές Κύριε Γκόμες θα κάνουμε ε, ηλεκτρονικό έλεγχο Πέρας 22-23 άρα απορρίπτεται 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 331 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Close. Adopted. Εγκρίνεται. 332. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 333. Ο πρόεδρος. υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 336 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Πέρασε ερασιωφορίες, 25-22 εγκρίνεται. Συμβαστική 12 νέα. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται 360 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ε, κύριε Μπρέντα, ψήφισατε δύο φορές νομίζω. Μάλιστα, καλά. Τελικά ψηφίζετε κατά, αλλά μία φορά. Συνεχίζει ο πρόεδρος, 361. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται η συμβαστική 15. 268. Υπέρ, κατά. Αποχές. Επαλήθευση λοιπόν και εδώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πρόκειται 368. Απεριθεί 18 υπέρ, 28 κατά. 371 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 377 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνω. Λέει ο πρόεδρος 378 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 379 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 381 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.83 υπέρ κατά επαλήθευση επαλήθευση τέλος Ψήφι 20 υπέρ 26 κατά. 384 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 385 <clears throat> υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 386 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 388 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 389 υπέρ κατά αποχές επανάληψη 389 υπέρ κατά επαλήθευση, επαλήθευση. Ορισμένοι μάλιστα ψήφισαν δυο φορές. «28 υπέρ 20 κατά εγκρίνεται». 390 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 391 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 392 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 59 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση τέλος 27 υπέρ, 21 κατά εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση λοιπόν κάπως.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 αποχές απορρίπτεται αυτή ε, του, της Επιτροπής ΔΕΒΕ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συνολικό ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος μα false λέει εδώ η εννέα, ε Άρα εκπίπτει αυτή. Λοιπόν, λειτουργική ψηφοφορία για το σύνολο, είπε ο Πρόεδρος. Mm. Τέλος της ψηφοφορίας. εγκρίνεται 33 ψήφοι υπέρ, μία αποχή και 14 ψήφοι κατά. Συγχαίρω την εισηγητρία. Θα συνεχίσουμε αμέσως για τη... Με συγχωρείτε, η Ενωτική Αριστερά επιθυμεί να λάβει το λόγο. Να ενημερώσω κύριε Πρόεδρε Συνεργούς ότι εμείς ως ΓΟΕ έχουμε κάποια μειοψηφία αρκετά σημαντική για την τροπολογία. Δεν έχει φτάσει ακόμη ο μεγάλος μουφτής, άρα θα αρχίσουμε τη ζήτηση για την, ε, την Ισία και αρχίζουμε μια μικρή εισήγηση. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Καστάλτο. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη πώς έχει η κατάσταση και το ότι λόγω των γεγονότων υπάρχουν αλλαγές στη μέση διάταξη. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, πρέπει να λάβουμε το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές και θα πρέπει όμως να είναι εδώ. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος η συζήτηση να είναι άσκοπη. Οπότε θα πρέπει να τους έχουμε εδώ. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε υπό αυτές τις ε, συνθήκες, λέει ο Καστάλντο, πρόεδρος. Ο πρόεδρος Μπρόκ. Να αναβάλουμε λοιπόν την συζήτηση περί την Ισίας για μετά το Πάσχα. Ή θα τα πείτε τώρα ή δεν θα τα πείτε καθόλου. Τι απόφαση λαμβάνετε. Αν δεν τα πείτε τώρα, δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση σήμερα ή πριν τις πασχαλινές διακοπές. Γιατί δεν διαθέτουμε απογευματινή συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε, κύριος, ε, σας είπα ότι δεν γίνεται ε, να το κάνουμε, αλλά έτσι όπως το λέτε, να, το κάνουμε. Όμως, από την άλλη μεριά, είναι μια χούφτα συνάδελφοι παρόντες. Καλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Οκ, okay, τότε αναβάλλεται, ματιώνεται για αυτή τη βδομάδα η συζήτηση για την Τινησία και βρίσκεται στην είσοδο του Κοινοβουλίου, στην κεντρική είσοδο, ο μεγάλος μουφτής. Σε μισό λεπτό θα πιει ένα καφεδάκι και θα έρθει. Πρώτα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Stay here, the Grand Mufti is in, he will be in a... Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι εδώ.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 ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι εδώ τον μεγάλο μουρτή της Αιγύπτου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Πιστεύω ότι η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας αποκτά έτσι ακόμα μεγαλύτερη σημασία δεδομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαμε τώρα τις πριν από λίγες ώρες. Εδώ δεν ε, σταβάζουμε βάζουμε το Ισλάμ συνολικά. 90% των θυμάτων εξάλλου των τρομοκρατικών Ισλαμικών επιθέσεων είναι μουσουλμάνοι. Άρα δεν πρόκειται εδώ πέρα να χωρίσουμε τους χριστιανούς από τους μουσουλμάνους. Χαίρομαι λοιπόν που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας. Ακριβώς περιμένουμε να μας μεταφέρετε τη θέση σας και να μας πείτε Πώς προτείνετε να συνεργαστούμε μεταξύ μας για να έχουμε ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς τρομοκρατία. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το μετήχουμε με συνεργασία μεταξύ μας. Έπειτα θέλω να υπενθυμίσω ότι τρεις μονοθεϊστικές ε, θρησκείες είναι θρησκείες ειρήνης και όχι θρησκείες πολέμου. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές και να διασφαλίσουμε την ειρήνη για τους πολίτες μας. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και σας ευχαριστούμε που ήρθατε κάτω από αυτές τις συνθήκες. στο όνομα ε, του Θεού, του Παντελεήμωνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας χαιρετίζω με τους χαιρετισμούς του Ισλάμ. Και οι χαιρετισμοί του Ισλάμ είναι η ειρήνη. Η ειρήνη σε σας, Η ειρήνη μην. Και για να, να αρχίσω, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου που με προσκαλέσατε εδώ και μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να μιλήσω μαζί σας για δεύτερη φορά μάλιστα. Πράγματι, ήμουν εδώ πριν από ένα χρόνο. Στιγμή που όλοι αντιμετωπίζουμε κοινέ προκλήσεις. Είναι προκλήσεις που μας υποχρεώνουν να ανοίξουμε διάβολους επικοινωνίας, διάλογο μεταξύ μας. Πριν λοιπόν περάσουμε στη συζήτηση μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποια σημεία, τα οποία ελπίζω ότι θα αποτελέσουν ε, πηγή εκκίνησης του σημερινού μας διαλόγου. Επιτρέψτε μου λοιπόν πρώτα απ' όλα να σας πω ότι για μένα ο κόσμος, ο ελεύθερος κόσμος καταδικάζει κατηγορηματικά χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία τα όσα έγιναν. Δεν καταφέρνουμε να βρούμε τις λέξεις, τα λόγια για να περιγράψουμε τις σημερινές τρομοκρατικές ενέργειες. Όλοι νιώθουμε δυστυχείς, ταραγμένοι και δυστυχώς δεν βρίσκω τα λόγια εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να εκφράσουν τα όσα αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Διότι η τρομοκρατία αυτή, η οποία χτύπησε σήμερα τις πόρτες μας, μας ε, βάλει όλους, όχι μόνο εμάς το Βέλγιο. Πριν από μερικές ημέρες, στην Αίγυπτο, επίσης η Αίγυπτος ήταν στόχος επίθεσης. 18 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο εξαιτίας της τρομοκρατίας αυτής. Η τρομοκρατία αυτή δεν γνωρίζει όρια, δεν γνωρίζει εθνικότητες, δεν γνωρίζει χώρες. Τα βάζει με όλους μας. Έτσι πλήττει την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αφρική και εξαπλώνεται παντού στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας και σήμερα ήρθε η στιγμή να δουλέψουμε μαζί, χέρι-χέρι. Και σήμερα είναι κατάλληλη στιγμή για να ανεώσουμε τη δέσμευση αυτή που έχουμε αναλάβει για συνεργασία και να πάψει να υπάρχει πια αυτό το φαινόμενο της τρομοκρατίας, να το διαλύσουμε, να το εξαρθρώσουμε. Σήμερα νιώθουμε όλοι δυστυχείς ξέροντας τι έγινε πριν από λίγες ώρες. Τι φταίνε τα θύματα αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ήμουνα στον Ταβός, στην οικονομική παγκόσμια διάσκεψη εκεί και μίλησα για αυτήν την κοινή ευθύνη που έχουμε όλοι μαζί και είπα ότι ο προφήτης λέει ειρήνη για όλους και αυτό ισχύει πράγματι για όλους, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό ακριβώς το μήνυμα του προφήτη για ειρήνη που απευθύνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο προφήτης έδωσε το παράδειγμα εκείνου του πλοίου πάνω στο οποίο βρισκόμαστε όλοι, ένα σκάφος. Όλοι λοιπόν βρισκόμαστε εκεί μέσα, οπότε δεν μπορούμε να δεχτούμε μία δράση, μία επίθεση η οποία θα βούλιαζε το πλοίο, γιατί θα βουλιάζαμε όλοι. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μαζί για να διασφαλιστεί η ακαιρότητα του σκάφους αυτού. Αυτό είναι το παράδειγμα λοιπόν που έδωσε ο προφήτης για να καταδείξει ότι αυτή είναι κοινή. Ζούμε όλοι σε αυτήν την ίδια γη που ανήκει σε όλους μας. Άρα οι προσπάθειες πρέπει να είναι κοινέ, συνδυασμένε για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Η Αίγυπτος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε όλα τα επίπεδα για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για να εξαρθρώσουμε αυτή την τρομοκρατία. Να το κάνουμε εμείς από την πλευρά των διανουμένων, των ε, κληρικών. Και όντως εμείς με το δικό μας τον τρόπο πολεμάμε για να εξαρθρωθούν οι βάσεις της τρομοκρατίας αυτής. Από την άλλη, θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου σε αυτά που είπε ο πρόεδρος πριν από λίγο, ότι δηλαδή τα γεγονότα αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζουν τις σχέσεις των μουσουλμάνων με τις άλλες κοινότητες, με τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Γιατί όλοι βρισκόμαστε σε αυτό το ίδιο πλοίο, όλοι μαζί. Η τρομοκρατία μα έκανε όλους θύματα και πολύ περισσότερο τους μουσουλμάνους από ό,τι τις άλλες κοινότητε, Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα βλέπουμε ότι η τρομοκρατία στις μουσουλμανικές χώρες είναι ακόμα πιο έντονη. Εκεί υπάρχουν τα περισσότερα θύματα, οπότε εμείς υποφέρουμε πάρα πολύ από τις τρομοκρατικές αυτές επιθέσει. Αυτό που είπε πριν ο πρόεδρο και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, όταν μελετάμε το Ισλάμ Και εγώ έχω μελετήσει και τις άλλες θρησκείες, την Μαγιαγραφή, ε, Παλαιά και Νέα Διαθήκη. Ε, λοιπόν, τα μηνύματα που έρχονται από αυτά τα Άγια Βιβλία, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι ότι καταδικάζουν την τρομοκρατία και ζητούν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ όλων μας. Τρίτον, εμείς ως κλήρικοι, έχουμε την ευθύνη να διαδώσουμε, να εξηγήσουμε την ε, καλή αυτή, την σωστή μορφή του Ισλάμ, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το Ισλάμ. Έτσι θα μπορέσουμε καλύτερα να συνεπάρξουμε και να συνεργαστούμε αμοιβαία. Ελπίζω ότι η σημερινή μας συνάντηση εδώ θα πάει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση και ότι θα ενισχύσει την ε, αντίληψη ότι βρισκόμαστε εδώ όλοι για να καταδικάσουμε την τρομοκρατία, να καταδικάσουμε αυτό που έγινε σήμερα και να καταδικάσουμε κάθε είδους τρομοκρατία όπου και αν λαμβάνει χώρα. Βρισκόμαστε εδώ ακριβώς για να διορθώσουμε, για να δώσουμε μια άλλη εικόνα του Ισλάμ σε σχέση με αυτά που έγιναν σήμερα. Ξέρετε ότι σήμερα ο κόσμος είναι θύμα αυτής της μάστιγας που είναι η τρομοκρατία. Επαναλαμβάνω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο πλοίο όλοι, το λέω και το ξαναλέω. Πρέπει λοιπόν να βοηθούμε ένα τον άλλο και να χρησιμοποιήσουμε από κοινού μέσα για να εξαρθρώσουμε αυτό το φαινόμενο. Να το εξαλείψουμε. Εγώ που είμαι επικεφαλής του Ντάρα Λιφτά, που είναι η ανώτατη αρχή, ξέρετε ότι η Φατφά είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπαγορεύσουμε κάποια πράγματα στο μουσουλμανικό κόσμο. Δυστυχώς όμως ορισμένοι χρησιμοποιούν με κακό τρόπο κάποια τέτοια κείμενα, δίνουν κάποια λαθασμένη ερμηνεία προκειμένου να επωφεληθούν οι ίδιοι. Τα χρησιμοποιούν προς όφελός τους, προς το δικό τους συμφέρον και για να δικαιολογήσουν αυτά που κάνουν σήμερα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν εξτρεμιστικές τάσεις με τις δικές του έννοιες, με τη δικιά του ερμηνεία και τις λαθεμένες ε, φατβά. Και έτσι έλεγα ότι η Ντάρα Λαφτά που είναι η ανώτατη θρησκευτική αρχή στην Αίγυπτο πολεμάει την τρομοκρατία αυτή από τη δικιά της την πλευρά. Και αυτό το κάνει δίνοντας ε, πραγματική ειλικρινή ερμηνεία των Αγίων Κειμένων προκειμένου να προστατεύσουμε τους νέους μας. Η Ντάρα Λεφτά, αυτή δηλαδή η ανώτατη θρησκευτική αρχή λοιπόν, αντελήθηκε το φαινόμενο και πήρε μέτρα από την αρχή, από πριν, για να προλάβει ακριβώς αυτόν τον ε, λαθεμένο λόγο της ΔΑΕΣ. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα παρατηρητήριο για να αντιμετωπίζουμε τις στραβές ερμηνείες του Κορανίου και προκειμένου να εξηγήσουμε τι ακριβώς λέει το Ισλάμ χρησιμοποιώντας την επιστήμη, τη σωστή ερμηνεία. Δημιουργήσαμε και ένα ειδικό κέντρο κατάρτισης μάλιστα το οποίο είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση της προπαγάνδας και αυτών των ε, λαθεμένων ιδεών και ερμηνεών. Το κάναμε. Και είναι ένας πυλώνας της λύσης αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Πιστεύουμε απόλυτα ότι αυτές οι ιδέες που μερικές φορές αγνούμε είναι μέρος της λύσης. Η Ντάρα Λιφτά χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες επικοινωνίας, χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα σε διάφορες γλώσσες μάλιστα, προκειμένου να έχει επαφές με πάρα πολύ κόσμο. Προκειμένου να μπορεί να έρχεται σε επαφή με όλους όσοι αναρωτιούνται και ψάχνουν απαντήσεις και να αντιμετωπίσουμε έτσι όλους αυτούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να δώσουν την λάθος ερμηνεία στο Ισλάμ. Έχουμε σελίδα Facebook, έχουμε και ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές σελίδες της Ντάρα Λεφτά που δημοσιεύει βίντεο σε 10 γλώσσες. Έχουμε επίσης και ηλεκτρονική σελίδα η οποία ονομάζεται «Η στο μικροσκόπιο». Η σελίδα αυτή λοιπόν που υπάρχει στα αραβικά και στα αγγλικά και στις δύο γλώσσες, ναι, υπάρχει. Και η σελίδα λοιπόν αυτή έχει ως στόχο να διορθώσει ακριβώς αυτές τις ε, λάθος έννοιες και τις λάθος ερμηνείες που δίνονται. Δημοσιεύσαμε μάλιστα και ένα, μια ηλεκτρονική εφημερίδα, σε ηλεκτρονική μορφή, στα αγγλικά. Η ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα που ονομάζεται Μπασίρα στα αραβικά, που σημαίνει ε, καλός τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Έχουμε μεταφράσει λοιπόν στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά χίλιες φατβά. Η μετάφραση αυτή των νομικών αυτών θρησκευτικών αποφάσεων έχει σαν στόχο να δώσει απαντήσεις και να αντιμετωπίσει όσα στραβά λέγονται από τις τρομοκρατικές ομάδες που βασίζονται σε λάθος ερμηνείες του Ισλάμ. Θέλω επίσης να πω ότι η σημερινή δικαιολογία για την τρομοκρατία στο μουσουλμανικό κόσμο και όχι μόνο. Οι δικαιολογίε που διαβάζουμε λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με τη διδασκαλία του Ισλάμ. Η διδασκαλία του Ισλάμ πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε τι μαθαίνουμε με επιστημονικό τρόπο και με λεπτομέρειες προκειμένου να υπάρξει απάντηση σε αυτή την απειλή για τον κόσμο ολόκληρο. Επιτρέψτε με εδώ να πω ότι το Ισλάμ το οποίο εμείς μάθαμε, που ήταν η βάση της εκπαίδευσής μας, είναι ένα Ισλάμ της ειρήνης. Είναι ένα Ισλάμ που μιλάει για την ελεημοσύνη, για την ανοχή και υπάρχει παράδοση από τον προφήτη που λέει ότι όσοι είναι ελεήμονες απέναντι στους άλλους θα δεχτούν ελεημοσύνη και από τους άλλους. Πρέπει δηλαδή όλοι και οι πιο ισχυροί να είναι ελεήμονες προς τους υπόλοιπους. Έτσι λέει ο προφήτης. Και το Κοράνι λέει ότι σας δημιουργήσαμε ε, άνθρωποι από έναν άνθρωπο και προκειμένου να ζείτε όλοι μαζί και να γνωρίζετε οι μεν τους δε. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι θρησκείες αποδέχονται την Θεία Δημιουργία. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν φτάνει να λέμε ότι το Ισλάμ είναι μια θρησκεία ειρήνης, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να παίρνουμε κατάλληλα μέτρα μέσω των ΦΑΤΦΑ για να δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορεί κανείς να δουλέψει για την ειρήνη. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικέ κοινότητες και είναι εκείνο της ε, αρχής. Ξέρετε ότι οι άλλες θρησκείες έχουν σημεία αναφοράς, έχουν δηλαδή συγκεκριμένες αρχές. Το Ισλάμ δεν έχει τέτοιες θρησκευτικέ αρχές. Ανθρώπους δηλαδή. Κάποιοι λοιπόν παριστάνουν ότι είναι η θρησκευτική αρχή του Ισλάμ. Κάτι το οποίο δεν ισχύει όμως στη θρησκεία του Ισλάμ. Έτσι άνοιξε η πόρτα στις στραβές εξτρεμιστικές ερμηνείες που δίνουν αυτές οι αρχές, που αυτοποκαλούνται αρχές του Ισλάμ. Όλοι μαζί πρέπει να καταπολεμήσουμε λοιπόν τους εξτρεμιστές αυτούς οι οποίοι από μόνοι τους πήραν αυτό το δικαίωμα να ερμηνεύουν τα κείμενα με στραβό τρόπο, με λαθασμένο τρόπο, χωρίς καμία απολύτως βάση το πραγματικό Ισλάμ. Στόχος των εξτρεμιστών αυτών, των τρομοκρατικών αυτών, είναι να διαδώσουν το χάος στον κόσμο. Όπως γνωρίζετε, η Αίγυπτος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή δύσκολη κατάσταση. Όλοι μαζί λοιπόν συνεργαζόμαστε προκειμένου να παρουσιάζουμε τη σωστή εκδοχή της συνύπαρξης και φτάνουμε στην ε, βάση και όχι να ακούμε αυτά που λέγονται δεξιά και αριστερά για να κρίνουμε το Ισλάμ. Η Αίγυπτος λοιπόν προσπαθεί σήμερα ε, με διαφάνεια, με πλήρη διαφάνεια να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση μετά από την εκλογή του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση πιστεύω. Ολονόν τα μάτια είναι στραμμένα στην Αίγυπτο ως την πηγή, την καρδιά της Μέσης Ανατολής. Μια χώρα που έχει πολύ σημαντικό ρόλο, κεντρικό ρόλο να παίξει σε περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ακριβώς εμείς ως Αιγύπτιοι πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτές του κόσμου. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την διεθνή κατάσταση, την διεθνή θέση της Αιγύπτου, κυρίως με την κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται. Ξέρετε επίσης ότι οι δημοκρατίες τουλάχιστον μία από τη βάση της δημοκρατίας ή τη διάκριση των εξουσιών. Η εκτελεστική, η νομοθετική, η εξουσία είναι διακριτές. Και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε και εμείς να υλοποιήσουμε, να το κάνουμε αυτό στη χώρα μας στην Αίγυπτο. Τέλος, θέλω να σας πω σε όλους σας ότι δεν υπάρχει καλύτερο όπλο κατά της άγνοιας, κατά του εξτρεμισμού παρά η καλή εκπαίδευση, η σωστή εκπαίδευση. Και είμαστε διατεθειμένοι εμείς ως ανώτατη θρησκευτική αρχή της Αιγύπτου, Νταρ αλιστά να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να εξηγήσουμε τις καλές, τις σωστές ε, φατφά, για να βοηθήσουμε και την περιοχή μας και το μουσουλμανικό κόσμο, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ε, πολιτισμού και θρησκείας για να καταλήξουμε στη συνύπαρξη. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ σε εσάς σήμερα. Ο Πρόεδρος. Uh, Ευχαριστούμε ε, πολύ. Εξοχότατε και Αντέλ Καριμαλάν, μεγάλη μου αυτή της Αιγύπτου που για άλλη μια φορά ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας απευθύνετε τους λόγους σας υπό αυτές τις τόσο εξωτικές ε, περιστάσεις και για την κατηγορηματική σας καταδίκη για τα όσα έγιναν εδώ στον ε, υπόγειο αλλά και στο αεροδρόμιο. Επίσης ε, νομίζω ότι λήφθη πάρα πολύ καλά το μήνυμά σας και αυτή η κάθε αντίθεσή σας στον ζωσπαστισμό και την τρομοκρατία. Έχουμε ένα σωρό συναδέλφους οι οποίοι τώρα θέλουν να κάνουμε μια συζήτηση οπότε πρώτα πρώτα λάβουν το λόγο αυτοί οι ευρωβουλευτές που θέλουν να μιλήσουν, να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις κατόπιν δε εσείς να έχετε το χρόνο, το περιθώριο να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλους μαζί οπότε πρώτα πρώτα ο κύριος ε, Πέτερλε από την Σλοβενία για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ, εδώ είμαι εξοχότατε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα πρώτα για αυτή την αλληλεγγύη που έχετε εκφράσει. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά στα οποία έχετε βοηθήσει μέσω του Ιδρύματος που αναφέρατε και συμφωνώ ότι η ειρήνη είναι στόχος, είναι αξία που διαπνέει όλες τις θρησκείες. Για πέστε μου, τι γίνεται όμως με εκείνους που καταχρώνται τις θρησκείες αυτοί δεν επιθυμούν διάλογο και ούτε βοηθούν σχετικά με δεν σας δεν βοηθούν την ε, τα λίφτα, το Ίδρυμά σας ε, σε σχέση με τον διαπολιτισμικό διάλογο όπως μας εξηγήσατε υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Ισλάμ και κάποιων άλλων θρησκειών οπότε και εγώ θεωρώ ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί μέσω του κόλπους του ιδίου του Ισλάμ και όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών θρησκειών. Πάντως θέλω να σας ερωτήσω, εσείς βλέπετε να υπάρχουν δυνατότητες, περιθώρια διαλόγου μεταξύ διαφορετικών ας πούμε πτερίγων και τάσεων στο Ισλάμ. Ευχαριστούμε Αλοίσια λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξοχότατε και σας ευχαριστούμε για τα όσα μας ε, είπατε, για όλα σας τα ενθαρρυντικά περί αλληλεγγύης. Εδώ, εδώ είμαι, εδώ είμαι, λέει η κυρία Γκίλ. Και θα ήθελα να σταθούμε στα εξής δύο σημεία. Πρώτα-πρώτα με προβληματίζουν τα σχετικά με την, την παράθεση αντιπαράθεση σε Σιητών. Αυτό μας ανησυχεί. Ε, νομίζω ότι η αντιπαλότητά τους γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Α, είδατε τι έγινε σε Ιεμένη, σε Ιράκ, σε Συρία. Και βέβαια, σε διάφορα μέρη στην Ευρώπη, οι δύο κοινότητες τα πάνε πάρα πολύ καλά. Όμως, πολλές φορές υπάρχει η εκμετάλλευση που σας ανέφερα. Εσείς τι, τι, βλέπετε, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το Ίδρυμά σας, μια που είναι βασικός θεσμός των Σουνιτών. Τι μπορεί να κάνει στον κόσμο τον Σουνιτικό, τόσο ώστε αυτό το χάσμα, αυτή η διαφορά να πάψει να γίνεται αντικείμενο χειραγώγησης και, και να συνεχίσει να υποδαβλίζεται αυτή η αντιπαλότητα. Επίσης, για πέστε μας, πώς θα μπορέσουμε να εξεφαλίσουμε το ότι η θέση των γυναικών και στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες θα βελτιωθεί. Πρόσφατα επισκέφθηκα τη χώρα σας, οπότε και προβληματίζομαι. Γιατί νομίζω ότι εκεί υπάρχει πισωγύρισμα όσον αφορά τη θέση και τον ρόλο των γυναικών, όσον αφορά τη συμμετοχή τους ε, ε, στα κοινωνικά κλπ. Και, και στην κοινωνία. Οπότε για το εκπαιδευτικό ίδρυμα σας πώς θα μπορέσει να αλλάξει την νοοτροπία σε σχέση με την θέση της γυναίκας. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος, δίνει τον λόγο στον επόμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά, λέει ο κύριος Γιούρεκ, που σήμερα λαμβάνω τον ε, λόγο στο Κοινοβούλιο. Ο, βεβαίως θα πρέπει να εκφράσω τη βαθιά μου αλληλεγγύη προς τις οικογένειες των θυμάτων για τις αποτρόπιες ε, πράξεις που σήμερα έλαβαν χώρα και θα συνεχίσω τώρα στη μητρική μου γλώσσα τα πολωνικά. Οπότε φορέστε τα ακουστικά σας για να παρακολουθήσετε την μετάφραση. Σήμερα θα ήθελα εξοχότατε να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι θετική η συνεισφορά της χώρας σας, γιατί πάντοτε υπάρχει τέτοια κατανόηση και πολλές φορές έχει γίνει κάτι τέτοιο ε, και έχουμε ε, ανταλλάξει τέτοιες θετικές απόψεις στο Κοινοβούλιο. Οπότε με τη σημερινή ευκαιρία σας παρακαλούμε να μας ε, βοηθήσετε και να κάνετε μία παρέμβαση για την υπόθεση αυτών των τριών νεαρών χριστιανών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση κάπου στην χώρα σας και συμπεριλαμβάνεται εκεί και ένας 15χρονος ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση σε κάποιο, κάποιο σοφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων γιατί ξέρετε τώρα οι χριστιανοί εορτάζουμε το Πάσχα πολύ σημαντικό αυτό και επίσης από ό,τι ξέρω μπορείτε να επηρεάσετε τα τεκτενόμενα στη χώρα σας και ε, επίσης απολαμβάνετε σεβασμού και όσον αφορά την ε, δικαιοσύνη. Οπότε θα ήμασταν ευγνώμονε αν κάνετε κάποια τέτοια χειρονομία πέρα αυτών των χριστιανών αυτή την εβδομάδα, την μεγάλη εβδομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο επόμενο ε, ο ο κύριος Παίρνουμε πρώτα-πρώτα να καταδικάσουμε αυτές τις ε, τρομακτικές επιθέσεις και ε, επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά θέλει να εκφράσει για τι οικογένειε των θυμάτων την ελεγγύη τη. Δεν πρόκειται αυτό να τελειώσει σήμερα εδώ. Οπότε και αυτό έχει σχέση με το συνεχιζόμενο το δικό μα έργο. Οπότε καλώ όρισε ο μεγάλο μοφτή αυτέ τι ώρε του πόνου που περνάμε και θέλω να σα πω ότι μας ε, ανησυχούν διάφορες πληροφορίες από την Αίγυπτο που φτάνουν όσον αφορά κάποιο είδους καταδίκε. καταδίκες. Ε, έχουμε πάρα πολύ βαριές ποινές που πέφτουν εκεί και στο Σινά υπάρχουν θέματα και εκεί πρέπει να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Θεωρούμε επομένω ότι δεν θα πρέπει όλα αυτά να μπερδευτούν ε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και οπότε δεν είναι δυνατόν για στο όνομα τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία να καταπατήσουμε όλα τα δικαιώματα. Οπότε για πέστε μας πώς προχωράνε τα πράγματα. Είναι δυνατόν να ε, έχουμε κάποια συνδιαλλαγή, κάποια συμφιλίωση και οπότε να ακούγονται όλες οι φωνές στην Αίγυπτο. Ε, ευχαριστούμε συνάδελφε Κούσο λέει ο, ο πρόεδρος. Έχει το λόγο κύριε Μπούχνερ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε με την διάθεση να συζητήσουμε για αυτό το ε, το θέμα σε τόσο δύσκολες περιστάσεις. Είπατε ότι όλες οι θρησκείες συμφωνούν ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερά. Ασφαλώς θα συμφωνείτε ότι δεν είναι και σωστό να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία με άλλη τρομοκρατία. Γι' αυτό ως υπάτη αρχή των μουσουλμάνων στην Αίγυπτο επιθυμώ να σε ρωτήσω συγκεκριμένα το εξής. Διαθέτεται την αυθεντία διαθέτεται και την εξουσία να εκδίδεται γνώμες για κάθε θανατική εκτέλεση. Συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό ισχύει και ενώπιον των ε, στρατοδικείων. Μιλώ για τους έξι οι οποίοι έχουν ε, καταδικαστεί σε θανατική ποινή ήδη από τον ε, περασμένο Μάρτιο για εγκλήματα τα οποία είναι αδύνατον να έχουν ε, εκτελέσει ήδη διότι ήταν ήδη στη φυλακή. Ήδη άνω των 500 ανθρώπων βρίσκονται υποκατηγορία και η ακρόασή τους κατά μέσον όρο ήταν της τάξης των 6 δευτερολέπτων ανακατηγορούμενο. Οι κατηγορούμενοι αυτοί εγκλείονται σε γυάλινα κλουβιά όπου δεν μπορούν καν να ακούσουν τα, τα τεκτενόμενα στην δίκη. Μπορείτε να εκδώσετε ε, γνώμες, πραγματογνωμοσύνες και για αυτές τις καταδίκες. Τρίτη ερώτηση. Στις φυλακές αποβιώνουν πολύ κρατούμενοι και λόγω της ελήψεως των απαραίτητων φροντίδων υγείας. Εκεί βεβαίως δεν μπορείτε να εκδώσετε ε, πραγματογνωμοσύνες. Μπορείτε να γύρετε την φωνή σας ως υπάτη ηθική αρχή στην ε, Αίγυπτο και την κατάστασή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούχνερ. Και τώρα κύριος Μπορκέτσι, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Εξοχότατε. Και εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για, και επίσης να στείλουμε την αλληλεγγύη μας σε ε, στα θύματα. Οπότε ε, τώρα έχουμε αυτούς τους ε, σφαγείς της ΆΕΣΕΣ που μέσα στο Πάσχα εκτελούν χριστιανούς. Βέβαια σα ευχαριστούμε για την καταδίκη προς εκείνα τα γεγονότα που έχετε εκφράσει αλλά και για τα σημερινά και πέραν αυτών εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ανώτατη ηγεσία της Ισλαμιστής Κοινότητας εδώ στις Βρυξέλλες και όπως είπατε τώρα έρθε η ώρα να καταδικάσουν και από αυτή τη θέση τα αυτά τα γεγονότα ε, οι Ισλαμικές αρχές και επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη την ευαισθησία που δείχνουμε για το αίμα χριστιανών το οποίο ε, χύνεται τώρα μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα λίγες μέρες πριν από το Πάσχα μας όπως είπε άλλος συνάδελφος. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Οπότε και σε σχέση με αυτό νομίζω ότι το σωστό είναι οι Ισλαμικές ε, αρχές να τοποθετηθούν όσον αφορά κάποιες ε, κυβερνήσεις. Να, Φερρυπίν για την Τουρκία η οποία έχει πάρα πολύ διφορούμενη στάση ως προς αυτούς τους ε, φερόμενους ως Ισλαμιστές που είναι ουσιαστικά τρομοκράτες και ουσιαστικά η Τουρκία ασκεί εμπορία. Εμπορεύεται το πετρέλαιο με αυτούς τους ανθρώπους. Τι λέτε, πώς βλέπετε αυτές τις κυβερνήσεις που στηρίζουν την δημοκρατία. Ευχαριστούμε κύριε Μπορκέτσιο, λέει ο πρόεδρος και τώρα η κυρία Καλνιέτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω εξοχότατε για το μήνυμά σας που ε, περιέκλει την ε, αηλενική αλλά και την καταδίκη ε, για τα γεγονότα αυτά και θυμάμαι ότι η μεγαλειώτης του ο βασιλεύς της Ιορδανίας είχε ομιλήσει στην Ολομήρια του Κοινοβουλίου και είχε πει ότι είναι κάθετα εναντίον της τρομοκρατίας και ότι η πιστοί του Ισλάμ είναι οι πρώτοι που θα επιλύσουν το πρόβλημα. Και για πέστε μας, αφού η πλειοψηφία των πιστών του Ισλάμ δεν μπορούν να κάνουν φωνή τους να ακουστεί. Και πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ε, λαμβάνει η χώρα από τις πρώτε τρομοκρατικέ επιθέσει και είχαμε και εκείνη την νεαρή Γαλλίδα η οποία κατόπιν των τραγικών γεγονότων των Παρισίων ε, είχε μέσω κοινωνικών δικτύων στείλει εκείνο το μήνυμα που έλεγε όχι ε, στο όνομά μου, όχι για λογαριασμό μου και πρόκειται για ε, πρωτοβουλία που προηγόταν από την Ισλαμική κοινότητα. Οπότε και σας ερωτώ Πώ βλέπετε εσεί τον ρόλο των θρησκευτικών ηγετών ούτως ώστε να υπάρχει πιο ενεργη, ενεργητική στάση συμπεριφορά τέλο πάντων των πιστών του Ισλάμ. Σάντρα, σε ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και δίνει το λόγο στην κυρία Γκόμες. Σε ευχαριστώ εξοχότατε που ήρθατε τέτοιες ώρες να μας επισκεφθείτε. Σας ευχαριστούμε και για όλα αυτά τα σοφά που μας αναφέρετε. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι τα περισσότερα θύματα της τρομοκρατίας είναι μουσουλμάνοι. Επίσης, μας είπατε για τον ρόλο σας, την αρμοδιότητά σας να ε, εκδίδετε αυτούς τους φετφάδες κατά του Ισλαμικού κράτους. Και είχαμε κάποιους ε, οι οποίοι είπαν ότι το Ισλαμικό κράτος έχει μπει και στα βίντεο παιχνίδια και εκμεταλλεύεται τους νέους που αισθάνονται αποξενωμένοι, που δεν έχουν δουλειά και ψάχνουν κάποια ευκαιρία. Να, τι συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη. Και οι επιθέσεις στην Ευρώπη, δεν ξέρω για σήμερα, αλλά οι άλλες ευρωπαϊκές επιθέσεις γίνανε από Ευρωπαίους. Αυτό θα πρέπει να μην το αγνοούμε. Ε, έχει να κάνει με τις δικές μας λάθος πολιτικές για το ότι δεν μπορέσαμε να προσφέρουμε στην νεολαία τις ευκαιρίες που προσδοκά. Οι ανισότητες, οι διακρίσεις κλπ. Βεβαίω όμως και οι θρησκευτικέ αρχές έχουν πάρα πολύ βαριές ευθύνες. Βεβαίω από την άλλη μεριά το μίσος δεν το προσβεύει καμία θρησκεία, ούτε το Ισλάβο, ούτε καμία, δεν πιστεύει στην τυφλιβία. Γι' αυτό και έρχομαι να σας ρωτήσω. Μίλησε ο συνάδελφος για το χάσμα, για την προστριβή σουνητών ε, σιητών, που πολλές φορές είναι η ρίζα του κακού ε, σε πολλά μέρη του κόσμου. Όμως υπάρχει χασμός και στους κόλπους των Σουνιτών, το είδαμε αυτό και στην Αίγυπτο αλλά και στην γειτονική σας ε, Λιβύη. Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία αλλά και τα Εμμυράτα ε, υποστηρίζουν μία παράταξη κατά άλλης. Επίσης και η Τουρκία και το Κατάρ. Να, για ποιο λόγο στην ίδια σας τη χώρα υπάρχουν προστριβές. Ε, βέβαια υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας γιατί θα πρέπει οι πολίτες να βλέπουν ότι οι ελευθερίες τις οποίες επιθυμούν υπάρχουν. Αλλιώς ξεσηκώνονται και ξεσηκώνονται κυρίως οι νέοι όπως ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν σε αυτή τη μαζική καταπάνωση των δρομινών δικαιωμάτων στην χώρα σας, στις διώξεις, στην καταστολή, κυρίως κατά των ε, νέων, των ζωντανών ανθρώπων που είδαμε πως ξεσηκώθηκαν στην πλατεία Τάρικ. Πέστε μας εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα. Τι γίνεται όσον αφορά το διχασμό στους κόλπους των Σουνιτών. Τι γίνεται όσον αφορά αυτή την ε, καταστολή που επικρατεί έχοντας ή δεν έχουν ε, μη έχοντες κάποια σχέση με τα θρησκευτικά πράγματα ε, αλλά εν πάση τόσο οδηγεί σε μη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας. Ο Πρόεδρος. Κύριε Αγκόμε, σας ευχαριστούμε. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στον συνάδελφο Σαφχάουζερ. Ευχαριστούμε. Εξοχότατε. Πρώτα πρώτα θέλω να σας πω ότι εκτιμούμε πάρα πολύ το τι γίνεται στη χώρα σας από τον πρόεδρο που δείχνει μεγάλο θάρρος και τότε που είχατε απευθύνει μια έκκληση ε, ούτω ώστε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, ε, προβληματισμός και είχαμε έναν θεολόγο και φιλόσοφο ε, τον οποίο ακολουθώ. Δηλαδή και εγώ ίδιος θέλω να σας πω ότι έχω υπερβολική στάση εναντί όλων των θρησκειών που λένε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και ο Θεός σας είναι μαζί μας. Αυτά απαντώνται σε πολλούς τομείς της πνευματικής ζωής και λέμε ότι τι γίνεται όταν περιμένουμε το Θεό, όταν θεωρούμε ότι ο Θεός ε, δεν είναι παρόν, ε, τότε κάτι λείπει από αυτό το δόμο, αυτή τη θρησκεία. Βεβαίω ε, και εγώ θαυμάζω τον Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και πέστε μας εσείς πώς λέτε τα πράγματα γιατί θυμηθείτε ότι στον Ιουδαϊκό κόσμο λένε ότι με τη βοήθεια του Θεού ε, θα τα καταφέρουμε ε, και ότι είναι μαζί τους ο Θεός αλλά εμείς ε, αυγούμε χαμένοι. Οπότε υπάρχει αυτή η υποταγή. Δηλαδή τι είναι εκεί που περιμένουμε ο Θεός ή δεν είναι. Ο Θεός βρίσκεται επί του Σταυρού. Κάτι το οποίο για πολλούς είναι απαράδεκτο. Όμως και αυτό είναι η αρχή της ελευθερίας, δηλαδή η αγάπη. Η αγάπη την οποία αρνηθήκαμε σε αυτόν τον Θεό μας. Οπότε για πέστε μας, εσείς πώς βλέπετε αυτού του είδους τον ρόλο του Θεού στο Ισλάμ, επίσης για πέστε μας για τον κοσμικό χαρακτήρα της κοινωνίας. Εμείς δίνουμε μάχη, αγωνιζόμαστε υπέρ αυτού. Περάσαμε από από διάφορες φάσεις και από τη φάση της αυτοκρατορικής διακυβέρνησης αλλά είναι κάποια βήματα πρόοδο οπότε ο κοσμικός χαρακτήρας της κοινωνίας θα πρέπει να σχετίζεται και με την πνευματικότητα άρα δηλαδή ο καθένας να έχει το ρόλο του δηλαδή να υπάρχει ο ρόλος της πνευματικότητας και ο ρόλος του κοσμικού χαρακτήρα της κοινωνίας και να υπάρχει κάποια διάκριση αλλιώς απουσιάζει η ελευθερία αυτό όμως δεν μας οδηγεί στο αντίθετο, ότι δηλαδή η πνευματικότητα ε, ότι δεν μπορεί να επηρεάσει θετικά. Όμως ο Θεός, ο δικός μας Θεός λέει ότι το δικό μου βασίλειο δεν είναι του κόσμου τούτου. Οπότε για πέστε μας για τον κοσμικό χαρακτήρα πώς τον βλέπετε, τι λέει το, το, το Ισλάμ, τι λέει για αυτά τα θέματα το Ισλάμ. Merci beaucoup pour ces questions euh, théologiques Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις θεολογικές απόψεις. Ο κύριος Μποστινάρα έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ με συγκινούν τα καλά σας λόγια. Εξοχότατε, ε, με μεγάλη μου ικανοποίηση συμμετέχω στην συνεδρίαση για ένα βασικό λόγο. Πρώτη φορά που άκουσα για την ανάγκη της αλλαγής της, της ε, Ισλαμικής σκέψης ήταν από τον Αιγύπτιο πρέσβη και χαίρομαι πολύ που είναι και ο ίδιος παρόν σήμερα. Σε αυτή τη τραγική στιγμή για τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη έχει έρθει η ώρα να εκφράσω και εγώ την αλληλεγγύη μου και να στείλω τα συλληπιτήριά μου στον Αιγυπτιακό λαό και στις οικογένειες οι οποίες ε, λαβώθηκαν τόσο βαριά από τόσες τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο αριθμός μεγαλώνει και δείχνει ξανά και ξανά ότι ο ίδιος ο μουσουλμανικός κόσμος είναι το πρώτο θύμα της νομοκρατίας. Τώρα δύο ερωτήσεις. Πρώτη. Η δέσμευση του Προέδρου Σίση να αλλάξει την ε, Ισλαμική σκέψη πώς μπορεί να υλοποιηθεί, πώς μπορεί να ε, εμπλέξει εντό εισαγωγικών και τους μουσουλμάνους ηγέτε. και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη μαζί σα, σε συνεργασία μαζί σα, για να αποφύγουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Μόλις επιστρέφω από την Ιερουσαλήμ και την Ραμαλά, όπου εντυπωσιάστηκα από την εικόνα που δίνουν οι δύο χώρες και οι σχολιαστές, οι όλοι, οι συνομιλητές μου όλοι, τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο της Αιγύπτου στην περιοχή αυτή ενώ η ίδια η χώρα αντιμετωπίζει τόσο μεγάλη τρομοκρατική απειλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρο. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε την λίστα των εγγεγραμμένων μελών, εκτός αν υπάρχει κανείς ακόμη. Αν συμφωνείτε, εξοχότατε, έχετε τη δυνατότητα τώρα να απαντήσετε με συνεκτικό τρόπο στις ερωτήσεις που τέθηκαν υπόψη σας από τους ε, συναδέλφους μου. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις αυτές πολύ σημαντικές και με βάθος που είναι ερωτήσεις που μας απασχολούν όλους και πράγματι θα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας μία προς μία. Σε ό,τι αφορά τον ε, ενδοϊσλαμικό διάλογο με τα διάφορα μέρη του Ισλάμ, δηλαδή αυτό τον εσωτερικό διάλογο του μουσουλμανικού κόσμου και του Ισλάμ. Βεβαίως ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Αυτό είναι και το νόημα της εκκλήσεώς μου, διότι η απομόνωση των διαφόρων μερών, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να διαλέγονται, το ένα μέρος να μην μπορεί να προσεγγίσει το άλλο, αυτή η απομόνωση μας οδηγεί στην σύγκρουση, είτε μεταξύ μουσουλμάνων, είτε μεταξύ μουσουλμάνων και άλλων. Ε, λαών ή άλλων ε, θρησκειών. Οι τρομοκρατικές ομάδες απεχθάνονται τον διάλογο. Οι τρομοκρατικές ομάδες έχουν την δική τους στρατηγική και το δικό τους σχεδιασμό τον οποίον προσπαθούν να εκτελέσουν με κάθε τρόπο. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτά να μπορέσουμε να οπλίσουμε τους νέους εντό εισαγωγικών, να τους θωρακίσουμε απέναντι σε αυτή την σκέψη. Γι' αυτό επιδιώκουμε τον διάλογο με τους νέους, για να τους εμποδίσουμε να προσελκύονται από αυτή την νοοτροπία της βίας. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να προσελκύσουμε τους νέους σε αυτόν τον διάλογο. Δυστυχώς όμως οι τρομοκρατικές ομάδες όσα έχουν κατορθώσει ως σήμερα αποτελούν πραγματικό καρκίνωμα, τα είπα αυτά και στον Ταβός. Καρκίνο που χρειάζεται αντιμετώπιση σε διάφορα στάδια. Πρώτα, πρέπει όπως είπα να θωρακίσουμε τους νέους απέναντι στην διάδοση αυτού του καρκίνου. Αυτή πρέπει να είναι η αρχή της θεραπείας. Αν η θεραπεία δεν αποδώσει αποτέλεσμα, πρέπει να αποκόψει κανείς το τμήμα εκείνο του σώματος το οποίο έχει πληγεί από τον καρκίνο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να θωρακιστούν οι άνθρωποι απέναντι σε αυτή την υπονομευτική ιδεολογία, με κάθε τρόπο. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που ακολούθησε σχετικά με τις εντάσεις μεταξύ Σιητών και Σουνιτών και όπου ναι, εντάσεις αυτές μεταξύ των δύο αυτών ομάδων μουσουλμάνων. Εδώ πρέπει να, γίνουν, γίνει κάποια, να γίνει μια διάκριση. Αφενός η πολιτική διάσταση του πράγματος που δεν μας αφορά. Γιατί αυτή είναι η υπόθεση των πολιτικών. Υπάρχει όμως και η άλλη διάσταση. Η θεολογική. Η θεολογική διάσταση, η θεολογική πτυχή των διαφορών μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εντάσεις. Ήδη από το 1940 στο Πανεπιστήμιο Ταλαζάρ Αλαζάρ, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε ακριβώς να εντοπιστούν οι ιδεολογικές διαφορές, εφόσον υπήρχαν να επιληθούν για να ε, ηρεμήσει ο διάλογος. Τώρα σε ό,τι αφορά το καθεστώς των γυναικών στην χώρα μας, είναι συνολικά το καθεστώς τους καλό, διότι το Αιγυπτιακό Σύνταγμα δεν προβαίνει σε διάκριση ή ουδήποτε είδους το κείμενο του ίδιου του συντάγματος δεν προβαίνει σε διάκριση ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα. Απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση βασισμένη στο φύλλο ή στο χρώμα του δέρματος και ούτε καθεξής. Αυτά τα λέει το Αιγυπτιακό Σύνταγμα, το οποίο απορρίπτει εντύπωτε διάκριση. Από την άλλη μεριά, οι γυναίκες στην Αίγυπτο ε, απολαμβάνουν μεγάλη ελευθερία εδώ και πολλά χρόνια. Άλλο σημαντικό γεγονό είναι ότι στην Αιγυπτιακή Βουλή συμμετέχουν πολλές γυναίκες και αυτό αποτελεί μια πρώτη στην Αίγυπτο. Εξάλλου, ε, σας επισημαίνω ότι σεβόμαστε τις γυναίκες και θέλουμε οι γυναίκες να χαίρουν του σεβασμού και με κανένα τρόπο δεν ζητούμε διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Αντιθέτως πάντοτε ταχθήκαμε υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή μάλιστα η έκκλησή μας έγινε ευνοϊκά δεκτή και στο πρόσφατα τροποποιηθέν σύνταγμα αλλά και στα προηγούμενα. σχετικά με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Καταβάλουμε πολλές και μεγάλες προσπάθειες και στην Αίγυπτο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το καθεστώς των χριστιανών στην Αίγυπτο ήταν πάντοτε ειδικό, ιδιαίτερο, με την έννοια ότι ποτέ δεν έχουμε προβεί σε οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, Αιγυπτιών χριστιανών. Οι Αιγύπτιοι χριστιανοί είναι Αιγύπτιοι πολίτες όπως οποιοδήποτε άλλος. Εγώ ο ίδιος προσωπικά έχω μεγαλώσει στην Αιγυπτική Ήπεθρο σε μια περιοχή όπου ε, ε, διαβιώνουν πολλοί χριστιανοί και ποτέ δεν αισθάνθηκα οποιαδήποτε διάκριση ή οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο αυτών πληθυσμιακών ομάδων. Να είστε λοιπόν βέβαιοι ότι αν υπάρχει ε, διάκριση αυτή ίσως προέρχεται από το παρελθόν αλλά δεν αρμόζει στον Αιγυπτιακό λαό και στην Αίγυπτο. Εξάλλου όταν η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται ενός προβλήματος ή μιας υποθέσεως, εμείς οφείλουμε να παραμείνουμε εκτός των δικαστικών αποφάσεων. Οφείλουμε να σεβόμαστε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να την αφήσουμε δηλαδή να κρίνει ανεξάρτητα τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν της. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και των σχέσεων ή μάλλον τον περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή της ελευθερίας στο όνομα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, από τη δική μας σκοπιά οφείλω να πω ότι η τρομοκρατία αποτελεί πρόβλημα που αξίζει δηλαδή που οφείλουμε να καταπολεμήσουμε με κάθε μέσον, διότι η τρομοκρατία μας απειλεί όλους, τους νέους μας, τις κοινωνίες μας, τους θεσμούς μας. Είναι λοιπόν δυνατόν έχοντας πει αυτά τα πράγματα να θεωρήσουμε ότι πρέπει να επιφυλάσσουμε μια φυσιολογική μεταχείριση απέναντι σε πρόσωπα που έχουν προβεί σε αυτές τις αποκρουστικές τρομοκρατικές πράξεις. Όχι, θα πρέπει να αυτούν ενώπιν τη δικαιοσύνης για να τους κρίνει. Και εν τέλει η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφανθεί. Εμείς ως θρησκευτικοί ηγέτες οφείλουμε να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Βεβαίως και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία ε, δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε όλες τις διαστάσεις και πτυχές τους. Ό,τι αφορά τις ε, καταδίκες σε θανατική ποινή. Οφείλω να σας πω ότι ε, αναφέρομαι σε αυτές που έχουν, τις αποφάσεις που έχουν εκδώσει τα στρατοδικεία. Τα στρατοδικεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Αιγυπτιακού δικανικού συστήματος. Τα δικαστήρια αυτά αποφαίνονται όπως και οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο. Ε, εντός των πλαισίων του νέου συντάγματος, όταν ένα στρατοδικείο ή και ε, πολιτικό δικαστήριο επιβάλλει την θανατική, θανατική ποινή, αυτή η θανατική θανατικη ποινη αυτη υποβάλλεται στον μουφτή της Αιγύπτου για να τοποθετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας νόμος Κανένας νόμος, σας βεβαιώνω. Δεν επιβάλλει την θανατική ποινή. Όχι, ας το πω διαφορετικά. Δεν υπάρχει κανένα σύνταγμα στον κόσμο που να μπορεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα των υποδίκων όπως το Σύνταγμα της Αιγύπτου, το οποίο ο Σύνταγμα της Αιγύπτου προσφέρει σημαντικότατες εγγύσεις πολύ περισσότερες από πολλές άλλες νομοθεσίες ανά τον κόσμο. Πριν λοιπόν να καταστεί αμετάκλητος η απόφαση, κάθε απόφαση των δικαστηρίων περνά από το φίλτρο διαφόρων επιτροπών, διαφόρων θεσμών, όπως είπα πριν να καταστεί αμετάκλητος και πριν να ε, ε, τεθεί υπόψη του Προέδρου της Δημοκρατίας εφόσον αυτό προβλέπεται. για αυτόν που ζήτησε καταδίκη των τρομοκρατικών αυτών επιθέσεων. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την έκκληση που ε, απίθυνε ο βασιλεύς της Ιορδανίας ό,τι αφορά την καταδίκη των τρομοκρατικών πράξεων. Κάθε δε μέτρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έχει την στήριξή μας. Στο Ντάριλ Φατβά έχουμε και διαδικτυακή πύλη σε διάφορες γλώσσες. Όπως λοιπόν η έκκληση που ε, διοχετεύτηκε στο διαδίκτυο από νεαρά Γαλλίδα μουσουλμάνα Πήραμε εμεί τον τίτλο για την ιστοσελίδα ε, μας. Διότι οι πράξεις αυτές είναι τρομοκρατικές πράξεις και δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την θρησκευτική σκέψη του Ισλάμ. Ο Νταέσ εξάλλου χρησιμοποιεί βιντεολήψεις αλλά χρησιμοποιεί επίσης και ναρκωτικά. Αυτά όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στα εγκλήματα που διαπράττει ο Νταέσου. Οι μαζικές δολοφονίες του Νταέσ. τα προπαγανδιστικά του βίντεο, το οργανωμένο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά οχριούν μπροστά τα βαριά εγκλήματα που διαπράττει. Άλλη ερώτηση που μου θέσατε αφορά την θέση της Αιγυπτιακής κυβερνήσεως για τους νέους Αιγυπτίους. Εδώ έχουν γίνει πολλά. Ο αριθμός των νέων μεταξύ των Αιγυπτίων βουλευτών έχει αυξηθεί. Και αυτό είναι μια πρώτη φορά στην ιστορία της Αιγυπτιακής Βουλής. Ο πρόεδρος Αλσισί όρισε το έτος 2016 ως έτος της νεότητας. σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν τρόποι για να συμβάλλουν στην προσπάθεια των νέων να επιδιώξουν τους στόχους τους και κάθε ε, κυβερνήτης επαρχίας στην Αίγυπτο ε, οφείλει να έχει και έναν ε, μεταξύ των προσωπικών συνεργατών του και έναν τουλάχιστον νέο σας ευχαριστώ και για όσα είπατε για τον πρόεδρό μας που μπορώ να σας βεβαιώσω ότι καταβάλει άοκνες προσπάθειες και ε, πολύ σημαντικές ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, για αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα, εγώ έχω να πω το εξή ότι ο παντοδύναμος Θεός έστειλε τους αγγελιοφόρους του για να διαδώσουν τον λόγο του και βεβαίω εάν κάθε πρόσωπο συμβάλλει στην υλοποίηση του Λόγου του Θεού, ο Θεός θα τον στηρίξει και δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ. Πρόκειται για μια φιλοσοφική πτυχή, όπως εξήγησατε και εσείς. Και εάν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τον Λόγο του Θεού, ο Θεός είναι κατά της ανατροπής. Και το Κοράνιο το ίδιο τα λέει αυτά. Έχει εκεί πολλές σεράτ που λέγουν απορρίψτε την ανατροπή. Τέτοια όπως βλέπετε και στην βίβλο και στην Καινή Διαθήκη. Το Ισλάμ δεν απευθύνει έκκληση για ανατροπές αλλά αντίθετα για οικοδόμηση, για αγάπη. Όπως το έχω πει και ξαναπεί, πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία με τον Λόγο του Θεού. Θέλουμε η δικαιοσύνη να καθιερωθεί, να βασιλεύσει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλη την ανθρωπότητα. Εάν πραγματικά ο λόγος του Θεού μας οδηγήσει σε αυτό το έσιον πέρας, ασφαλώς εμείς ε, θα είμαστε διευτυχέστεροι. Δεν θυμούμε πλέον ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της ερωτήσεως σας, αλλά ε, ήταν ε, συνολικά για την Αίγυπτο και πάντως σας ευχαριστώ για την στήριξη που προσφέρετε στην Αίγυπτο και που δηλώσατε ότι κατανοείτε την δυσχέρεια των περιστάσεων που ζει η Αίγυπτος. Και ε, επιβεβαιώνω τα όσα είπατε πράγματι, ο μουσουλμανικός κόσμος στο σύνολό του υποφέρει, πάσχει, ολόκληρος ο κόσμος, διότι η δυστυχία δεν έχει σύνορα. Μας πλήττει όλους. Και αυτό απαιτεί λοιπόν να φανούμε όλοι αλληλέγγυοι και να συνεργαστούμε για να αγωνιστούμε κατά, να, ε, Ο δε πρόεδρος μας Αλσισί ε, έχει δεσμευτεί στην κατεύθυνση αυτή. Θέλει την διατήρηση του κράτους δικαίου και επιθυμεί ταυτόχρονα να διατηρήσει με ξεκάθαρο τρόπο την διάκριση των εξουσιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Your Ευχαριστούμε πολύ εξοχότατε μεγάλη μου της Αιγύπτου. Ε, Καρή Μαλάμ, πάρα πολύ ενθαρρυντικά και ξεκάθαρα τα όσα μας εξηγήσατε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και επίσης ε, στο ίδιο μικρό σχήματο κινήθηκε και ο πρόεδρο μα ο κύριο Μπρόκ, ο οποίο στο Κάιρο είχε συναντήσει πρόσφατα με τι Αιγυπτιακέ Αρχέ. Σα ευχαριστούμε για την επίσκεψή σα είναι απίστευτο το όσα σήμερα, αλλά και τραγικά ε, ε, και για το Βέλγιο, αλλά και για τα θεσμικά όργανα. Οπότε όσα είπατε και η καταδίκη της τρομοκρατίας από πλευρά σας έχουν ακόμα πιο μεγάλη σημασία και σας ευχαριστούμε. Σε δύο λεπτά, λέει ο Πρόεδρος, θα συνεχίσουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης. Dear colleagues, we shall continue with our... Συνεχίζουμε, συναδελφοί, τη συνεδρίασή μας. Έχουμε το θέμα του αστυμών 11 διατάξεως, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης, τον κύριο Ριάντ Αλμαλκή. Η εξοχώρηση του μας ετοίμησε με την παρουσία του σήμερα στο Κοινοβούλιο. Ο κ. Αλμαλκή επί Μακρόν διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών. Σήμερα, εξοχότατε ήρθατε στις Βρυξέλλες, μία μέρα μεγάλης τραγωδίας. Τα γεγονότα του αεροδρομίου Ζάβεντεμ και του σταθμού του υπόγειου του Μάλμπεκ εδώ κοντά. Καταδικάζουμε την ε, τρομοκρατική αυτή επίθεση και έχουμε παρακολουθήσει τη διαδικασία στην ε, Εγγύης Ανατολή και θέλουμε επίση τη δική σα γνώμη, τη δική σα ανάλυση για το πώ έχουν σήμερα τα πράγματα και τι μπορούμε να περιμένουμε τους αμέσως επόμενου μήνε. Ενδεχομένω, ίσω θα μπορούσατε να μα ενημερώσετε ελαφρώς για τι δικέ σα απόψει όσον αφορά την πρόσφατη γαλλική πρωτοβουλία αλλά και επίση την ε, φιλόδοξη προσπάθεια τη επανέναρξη τη συνεχής διαδικασία από πλευρά Κοινοβουλέου. Ήταν χρήσιμο να ακούσουμε πώ έχουν προχωρήσει τα πράγματα, πώ έχουν τα πράγματα όσον αφορά ε, τις διαδικασίες ε, συνδιαλλαγής στην Παλαιστίνη, ε, στην Παλαιστίνη αλλά και ευρύτερα στην ε, περιοχή Κίνης, πες μας γνώμησες για το Ιράκ, για τα γεγονότα και στην Βόρειο Αφρική. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, επιτρέψτε να σας πω για το ότι καταδικάζουμε τέτοιες τρομοκρατικές ε, απόπειρες όπως έγιναν εδώ στις Βρυξέλλες. Και ξέρετε ότι η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε εθνικότητα, ούτε πατρίδα. Οπότε όλοι από κοινού θα πρέπει να δώσουμε αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας όπου χτυπά και θα πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, απειλή και θα πρέπει να την εξαλείψουμε εντελώς συμφωνώ μαζί σας ότι πέραν της καταδίκης θα πρέπει να απευθύνουμε τα συλληπιτήρια. προς τις ε, οικογένειες των θυμάτων και επίσης να ευχαριστούμε περαστικά στους ε, τραυματίες. Με μεγάλη με σήμερα απευθύνουμε στην Επιτροπή σας η οποία έχει τέτοιο κύρος και έχω μήνυμα ειρήνης. Ήρθε η ώρα ούτως ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε ένα τέλος ε, στην πιο μακροχρόνια κατοχή της ε, σήμερα. Θα ξέρετε τι συμβαίνει στην ε, Παλαιστίνη. Κάθε μέρα υποφέρει εκεί ο κόσμος και κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι δυνατόν να επισκιαστεί από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή γιατί η Παλαιστίνη είναι το κλειδί για ειρήνη και ασφάλεια όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε όλο τον κόσμο και άπαξ και αυτή η σύγκρουση δεν έρεται θα έχουμε τις εξτρεμιστικές ενέργειες και θα στρατολογούν ε, αυτοί οι τρομοκράτες. Οπότε εμείς θέλουμε να υπάρξει μια πραγματική ειρήνη, να είναι βάση το διεθνές δίκαιο και οι επιταγές του κράτους δικαίου. Και από τότε που υπερογράφηκε η συνθήκη και η συμφωνία του Όσλο με κάθε ευκαιρία καταγγέλουμε την κατοχή και προωθούμε την ε, λύση των δύο κρατών ε, σε συνεννόηση με το κράτος του Ισραήλ. Δυστυχώς ε, το μόνο το οποίο είχαμε ήταν περισσότερους επικισμούς, κατάτμιση της κατάστασης ε, περισσότερες ε, ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν κυρίες και κύριοι παρά όλες αυτές τις δυσκολίες ο λαός μας έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα έδειξε την θέληση όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον και ξέρω ότι τα μέσα ενημέρωσης σας δείχνουν την απελπισία και τον θάνατο από τη χώρα μου αλλά ε, επιτρέψτε μου τώρα να σας δείξω ε, το, να σας εξηγήσω πώς κάποιοι Παλαιστίνοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουμε μεγάλη θέληση. Η κυρία Χανάν Αλμόρ ε, ήταν ε, μία δασκάλα που έδειξε πάρα πολύ αφοσίωση και αποφασιστικότητα και έλαβε το βραβείο του, του καλύτερου δάσκαλου. Προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει ότι οι μέλους τη γενιά θα πρέπει να, να, έχουν το ίδιο πνεύμα. Επίσης, άλλο δείγμα αριστείας, ο Μπαράχ Σαράρι, ο οποίος είναι 8 ετών και μένει στο Αλχέλβε που είναι ένας καταβλισμός προσφύγων στον ε, Λίβανο και ε, μετά από κάποια διαδικασία προαπλασιασμών απέδειξε ένα θεώρημα μαθηματικό ε, χωρίς υπολογιστή, χωρίς αριθμομηχανή και δοκιμάστηκε η απόδειξή του από Άγγλους, Γάλλους και άλλους επιστήμονες και θεωρήθηκε και πήρε το βραβείο του πιο νέου μαθηματικού στον κόσμο. Να ένα παράδειγμα προς μίμηση πρέπει να το μιμηθούμε όλοι εμείς που ζούμε στην ε, κατοχή. Ε, να, ε, πώς είναι δυνατόν να αποδείξει κανείς ότι αξίζει την ανεξαρτησία και την ελευθερία. Όμως το Ισραήλ συνεχίζει να καταπατά τα όσα έχουν συμφωνηθεί ε, να μην σέβεται την λύση των δύο κρατών. Θα πρέπει να βρεθεί μια πρακτική λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετηθεί όσον αφορά τους Ισραηλινούς επικισμούς, αλλά, αλλά δεν αρκεί τούτο το Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνει από λόγια. Οπότε και θα πρέπει ε, τα λόγια να γίνουν έργα. Επομένως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς δεν ωφελείται από αυτή την κατοχή. Έχουμε ε, τις κατευθυντήρες γραμμές, έχουμε τα διαβήματα που θα πρέπει να αναλάβουμε και δυστυχώς ε, ε, κάποιες πλευρές χρησιμοποιούν όλα αυτά ούτως ώστε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα και προσπαθούν να δουν το πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι επικισμοί από, κάποιες, από κάποιους κύκλους επιχειρηματικός. Δεν θα πρέπει επομένως η Ευρώπη να πέσει θύμα ε, και ούτε θα πρέπει πια να συνεχίσουμε κάποιο μποϊκοτάρισμα αυτής της διαδικασίας κατά του Ισραήλ. Όχι, να μποϊκοτάρουμε τους επικισμούς αλλά όχι το καθεαυτό το κράτος του Ισραήλ. Επομένως ε, όλα αυτά βλέπετε το πόσο μας έχουν επηρεάσει. Έχουμε αυτή την κατάτμιση της ε, χώρας, αυτούς τους επικισμούς βλέπουμε ότι μας έχουν αποστερήσει το εισόδημα και έτσι καταργείται στην πράξη η λύση των δύο κρατών. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, Παλαιστίνη. Ε, θεωρείται κατηγορίας ε, γάμα όσον αφορά τις αναπτυξιακές δυνατότητες γιατί πρόκειται για το 61% της χώρας μας αλλά έχουμε τις επιχειρήσεις αλλά και την κυβέρνηση του Ισραήλ που πανεμποδίζουν κάθε μας τέτοια προσπάθεια και επίσης δυναμητίζουν τα έργα και προγράμματα που ξεκινάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των ε, σχολείων που προσπαθούν να καλύψουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες του λαού μας. Έχουμε κάποιες προσπάθειες ε, τέτοιες ε, σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο οι δανειοδότες οι εσείς. Όμως παρόλα αυτά το Ισραήλ τίποτα από αυτά δεν σέβεται κυρίες και κύριοι το Παλαιστινιακό κράτος διψά για την απελευθέρωση θα σταματήσει αυτή η κατάσταση της ε, εχμαλωσίας, της υποταγής του λαού. Θα πρέπει και εμείς να μπούμε ως ίσοι στην κοινότητα των εθνών και να αποκτήσουμε αυτονομία, κυριαρχία στο ε, πρωτεύουσα παραμείνει ε, το ε, να γίνει μάλλον η Ιερουσαλήμ όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ειρηνικούς τρόπους έτσι να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας και θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα ούτω ώστε να προωθηθούν κάποιες βιώσιμες λύσεις για την ρύθμιση των δύο κρατών δεν θα πρέπει να είμαστε σε ομοιρία δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια δύναμη κατοχής όχι σε όλα αυτά. Δεν θα πρέπει ο κόσμος να συνεχίσει να είναι μάρτυρας μιας τέτοιας κατοχής. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει τόση καταστροφή, να υποφέρουμε τόσο πολύ. Άρα είναι ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει αυτούς που υποφέρουν από αυτή την κατοχή. Βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε πώς το Ισραήλ καταπατά το διεθνές δίκαιο. Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Αυτό που θέλουμε είναι μια πολυμερή λύση και έτσι να προστατευτεί και να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών και έτσι να μπορέσουμε να εγκαθιδρύσουμε ένα παλαισθηνιακό κράτος σε στενή συνεργασία με τους Γάλλους φίλους, ούτως ώστε να προωθηθεί αυτή η λύση μιας διεθνούς ειρηνευτικής διασκέψεως θα πρέπει με αυτή την διάσκεψη να ορίσουμε κάποιες παραμέτρους των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Οπότε να οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ξεκάθαρο και κάποιους ούτως είπεν κανόνες παιχνιδιού που θα σεβαστούν και οι δύο πλευρές υπέρ της λύσης των δύο κρατών, υπέρ του τέλους του επικισμού. Αλλά βέβαια δεν είναι δυνατόν να στηριχθούμε ε, στην καλοπιστία, στην καλή θέληση της Ισραηλινής κυβέρνηση και κυρίως της σημερινής κυβέρνηση, που έχει δείξει ότι δεν σκέφτεται καρφάκι για την ε, λήξη της κατοχής. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στο διεθνές δίκαιο ε, όπως ας πούμε την κρίση του Ιράν που εγνώρισαν ειρηνική λύση και όχι μια μεγάλη σύγκρουση. Άρα μπορούμε έτσι να έχουμε κάποια, ε, κάποιο διεθνή φορέα. Και έτσι και ε, στις 18 Ιανουαρίου του 2016 είχαμε μια συνάντηση πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι έχει φανεί πόσο ενδιαφέρεται στα σοβαρά η κοινότητα να βάλει ένα τέλος στην ε, κατοχή της Παλαιστίνης. Εδώ και σήμερα κυρίε και κύριοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μια εκστρατεία, εκστρατεία που είναι κατά της ύπαρξης του έθνους μας και είδαμε την κλιμάκωση της βίας των ε, επικιστών και τους βοηθά βέβαια ο Ισραηλινός στρατός. Θεωρούν ότι μπορούν να καταστρέφουν σπίτια και τζαμιά ατιμωρητή. Υπάρχει με αυτή η εκστρατεία του μίσους της Ισραηλινής κυβέρνησης. Τελούμε υπό συνεχείς επιθέσεις και απειλές. Και δεν αισθανόμαστε ασφάλεια ούτε καν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου η διεθνής προστασία είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να υπάρξει. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την παράταση της σημερινής κατάστασης που μπορεί να κλιμακωθεί σε ένα ολοκληρωτικό χάος ανεξέλεγκτο με ανυπολόγιστες συνέπειες. Θυμάστε ε, το, το πώς πυρπολήθηκε η οικογένεια Γουάμψη όταν τους, τους επιτέθηκαν στο ίδιο του το σπίτι. Ε, αυτοί που επιτέθηκαν αλλά και οι υποστηρικτές τους είναι ατιμόρυτοι, έτσι νομίζουν ότι είναι. Και πριν από τρεις ε, μέρες αποφάσισαν να ε, κάψουν τους μάρτυρες των αποτρόπιων πράξεων τους που έκαψαν επομένως το πυρπόλησαν με εμπρισμό στο σπίτι του τον μοναδικό μάρτυρα και την οικογένειά του. Οπότε θα πρέπει να δούμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε συμβάλει τις απόψεις σε διαφορετικά επίπεδα και αυτές οι φρικαλαιότητες, αυτές οι δυσκολίες, τα βάσανα, τα καθημερινά είναι σε βαθμό πάρα πολύ έντονο και για να τα καταφέρει κανείς, να τα καταλάβει θα πρέπει να τα περάσει ο ίδιος οπότε θα πρέπει επομένω να συνεχίσετε να επισκέπτεστε την Παλαιστίνη σας καλό όλοι όποτε σας εξυπηρετεί. Ελάτε και να δείτε την αλήθεια με τα ίδια σας τα μάτια. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό κανείς να γίνεται μάρτυρας ε, των γεγονότων και να μπορεί έτσι να αναλάβει φράση αγαπητοί φίλοι. Εν κατακλείδη, σας επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είπα στην αρχή. Απερίφραστη καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων και συλληπιτήρια προς τα θύματα αυτών. Και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Υπουργέ, φυσικά είναι έκτακτες οι συνθήκες σήμερα. Γι' αυτό και έχουμε πολύ λιγότερους παρόντες εδώ από ό,τι κανονικά, σε μια κανονική συνεδρίαση. Πάντως σίγουρα θα υπάρξουν αρκετά σχόλια. Κύριε Αναγκόμες έχει πρώτα το λόγο εκ μέρους των σοσιαλιστών, από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήρθετε και που καταδικάζετε τις τρομοκρατικές ενέργειες. Φαίνεται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στον κόσμο ολόκληρο και στη δικιά σας περιοχή να γίνεται κάτι συνηθισμένο, αλλά εμείς αυτό το απορρίπτουμε, το καταδικάζουμε και αυτό που είπατε εσείς ήταν πολύ σημαντικά. Επίσης ευχαριστούμε που μας λέτε ότι οι συζητήσεις για την ειρήνη στην Παλαιστίνη και ανάμεσα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ είναι μια άρνηση στα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα επιθέσεις δηλαδή. Είναι κάτι λοιπόν που και εμείς καταδικάζουμε και απορρίπτουμε για όλους. Είναι κρίμα που δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί δεν έχουν υλοποιηθεί στη συνέχεια. Η ερώτησή μου είναι εξή. Τι μπορείτε να μας πείτε για τη διάσκεψη αυτή που ετοιμάζεται στο Παρίσι. Δεν πρόκειται μόνο για το Παρίσι, πρόκειται για την ίδια την Ευρώπη. Πού βρίσκεται αυτή η Ευρώπη η γαλλική κυβέρνηση δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν χρειαζόμαστε μόνο τη γαλλική κυβέρνηση, χρειαζόμαστε την Ευρώπη να είναι παρούσα εκεί. Η Ευρώπη πρέπει να δεσμευτεί για να σταματήσει η κατοχή της Παλαιστίνης. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες για την εμπλοκή της Ευρώπης αυτό και μπορείτε να μας πείτε η ενότητα του λαού της Παλαιστίνης. σε σχέση με τα όσα γίνονται στη Γάζα. Μπορείτε επίσης να μας πείτε τι κάνει η κυβέρνησή σας προκειμένου να καταπολεμήσει την αντίληψη που επικρατεί όσο γίνεται όσο περνώ ο όλο και περισσότερο μεταξύ των μορφωμένων Παλαιστινίων. που δείχνουν απελπισμένοι όσον αφορά το Παλαιστινιακό κράτος και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τους κανόνες και από πλευρά του ελληνού κράτους και τελικά φοβούνται ότι υπονομεύεται η θέση αυτή για τα δύο κράτη. Και εσείς το βλέπετε έτσι. Αν όντω υπάρχει αυτή η απελπισία μεταξύ των μορφωμένων Παλαιστινίων, αυτό θα έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για την επίτευξη του στόχου. Πώς βλέπετε εσείς το τέλος αυτής της κατοχής, το κράτος της Παλαιστίνης δηλαδή, πώς το βλέπει και πώς προχωράει σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το κράτος σας απέναντι στα διεθνή φόρα. Ευχαριστούμε κύριο Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Επιτρέψτε μου να σας θέσω υπόψη το εξής. Η άρνηση της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Βεβαίως έχω να πω το εξής. Κάθε έθνος, κάθε λαός έχει το δικαίωμα να εκλέξει την κυβέρνηση που επιθυμεί. Όμως και οι άλλε χώρε, οι άλλοι λαοί έχουν το δικαίωμα να κρίνουν τα πεπραγμένα της κυβέρνηση αυτή. Η κυβέρνησή σα ασκεί πραγματικά εξουσία στη λωρίδα της Γάζας ή έχει η λωρίδα της Γάζας πια τη δική της γνώμη. Πώς είναι η σχέση της κυβέρνηση όσο με τη χαμά. Και κάτι ακόμα επιθυμώ να θίξω. πώς ορίζεται σήμερα την θέση των Παλαιστινίων. Για το Ισραήλ, ποια είναι η θέση των Παλαιστινίων απέναντι στο Ισραηλινό κράτος. Σας ευχαριστώ κύριε Κιωρέκ. Η κυρία Σακοράφ. Κύριε Μάλικη, το 1993 η λόγια και στη συνέχεια η Παλαιστινιακή Αρχή αναγνώρισαν το τα σύνορα του Ισραήλ ε, στα σύνορα του το 1996 μια πανηγυρική συνέλευση της, Πανε... της Παλαιστινιακής στη Γάζα, παρουσία του κυρίου Κλίντον, αφαιρέθηκε από την Παλαιστινιακή διακήρυξη οποιαδήποτε αναφορά στην καταστροφή του Ισραήλ. Αντίθετα μέχρι σήμερα, το Ισραήλ όχι μόνο αρνείται να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, αλλά δεν αναγνωρίζει ούτε καν τα δικά του σύνορα. Μόλι τον προηγούμενο μήνα, μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα, ρώτησα τον πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνα τη ΝΕΣΕ, τον κύριο Χάνινγκπιν, να μα πει ποια είναι τα σύνορα του Ισραήλ και φυσικά δεν μα απάντησε. Αυτονόητο μου φαίνεται αφού το Ισραήλ συνεχίζει να προσαρτά παλαιστινιακά εδάφια ακόμη και τώρα, με τελευταία 2.500 τρέματα τη πιο εφορή περιοχή στον Ιορδάνη, συνεχίζοντα να επικίζει την περιοχή και τη δυτική όχη, όχθη, αγνώντα και παραβιάζοντα για μια ακόμη φορά το διεθνέ δίκαιο, τι καταδικαστικέ αποφάσει των διεθνών οργανισμών και του Διεθνού Δικαστηρίου τη Χάγη. Και δεν μπορώ να μην επισημάνω βεβαίω και την δήλωση του κυρίου Νατανιάχου που θέτει σε κίνδυνο οποιαδήποτε εφικτή λύση και για τα δύο κράτη, που λέει ότι γκρέμισε τι έξι χρηματοδοτούμενε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπιστικέ δομέ επειδή κατασκευάζεται, όπω ο ίδιο ισχυρίζεται, κατασκευάστηκαν παράνομα. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τολμάει, να, κατά τη δική μου άποψη, να προβάλλει την παραμικρή αντίδραση απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη πολιτική, ακόμα και όταν αναγκάζεται να πάρει μέτρα όπω είναι αυτά των, τη σήμανση των προϊόντων από του παράνομου Ισραηλινού επικισμού. Και συμφέρει φυσικά μέσω τη κυρία Μαγκερίνη να δηλώσει ότι δεν, η οποία δηλώνει δεν υποστηρίζει με κανέναν τρόπο τον μποϊκοτάζ των Ισραηλινών προϊόντων διαβεβαιώνοντά τον ότι η ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων αυτών αφορά καθαρά το κάθε κράτο ξεχωριστά. Σα ρωτάω λοιπόν, ποιο νόημα έχουν οι συμφωνίε που έχετε υπογράψει, αφού είστε οι μόνοι που δεσμεύεστε από αυτέ. Τι βάρο έχουν οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν είναι δεσμευτικέ για τα κράτη-μέλη και δεν έχουν το χαρακτήρα κυρώσεων κατά του Ισραήλ. Και η τελευταία μου ερώτηση, τι άμεσο και συγκεκριμένο ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει αποτέλεσμα και να μην είναι υποκριτικά ευχολόγια. Αυτό και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σακοράφα. Ο κύριος Μπούχνερ έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που υπό τι ε, δυσχερεί αυτές τις περιστάσεις προσήλθατε σήμερα ενώπιον μας. Ευχαριστώ και για την ευγενή σας πρόσκληση για την διεξαγωγή επισκέψεως. Ήδη πέρσι είχαμε έλθει να σας δούμε και πολύ απολαύσαμε την φιλοξενία σας. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη. Υπάρχουν αναφορές στον τύπο που λένε ότι σύντομα θα διεξαχθεί νέα συνάντηση μεταξύ Χαμάς και Φατάχ στην Τόχα μπορείτε να πείτε λεπτομέρειες σχετικά και ιδίω βλέπετε κάποια πιθανότητα, κάποιο ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια προσέγγιση ή κάποια συνεννόηση που ε, θα ήταν βεβαίως ε, πάρα πολύ ευεργετική για ολόκληρη την περιοχή σας. Δεύτερη ερώτηση. Η συμφωνία για τις αεροπορικές συγκοινωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ισραήλ που συνήθει πρόσφατα και που φαίνεται πως έγινε ε, το λάθος να μην περιληφθεί η Παλαιστίνη όπως θα θέλαμε εμείς. Μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Μπορείτε να μας δώσετε εξειδικευμένες συμβουλές για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε συγκεκριμένα στο θέμα αυτό. Ο κύριος Μποστινάρου, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Πραγματική είναι, είναι γνήσια χαρά μου που σας ξαναβλέπω. Μόλις επέστρεψα από Ιερουσαλήμ και Ραμαλά την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Μιλήσατε για την γαλλική πρωτοβουλία, ορισμένη από τους συναδέλφους μου ζητούν την εκτίμησή σας για τα επόμενα βήματα. Έχω δύο ερωτήσεις τώρα πιο συγκεκριμένες. Πρώτο, σχετικά με, τη, με το ενδεχόμενο κυβέρνηση τη Εθνικής Ενότητας στη Ραμαλάχ για όλους τους Παλαιστινίους που θα αναλάβει τα Ινία και θα διακυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας. Δεύτερο, η επίσκεψη τη Χαμά στο Κάιρο και οι διαπραγματεύσει με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Έχετε περισσότερα να ε, πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πουστινάρο. Ο κύριο Λίτς. Ευχαριστώ που ήλθατε διακόπτη. Να ξαναρχίσω γιατί ίσως δεν ακούσατε την αρχή της παρεμβάσεώς μου. Ευχαριστώ που ήρθατε ειδικά σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες να μας δείτε και που δείχνει πόσο πολύτιμη είναι η ελευθερία και η ειρήνη που τόσο πολύ συγκλονίστηκαν σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και που μας δίνουν και μια γεύση από το τι ζείτε εσείς στη δική σας περιοχή είμαστε στο πλευρό σας για την αναζήτηση της λύσης των δύο κρατών και μακάρι να επιτύχετε και εθνική ενότητα ε, στην πολιτική σας υπέρ όλων των Παλαιστινίων. Έχουμε την πληροφορία ότι πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη στην ηγεσία της Φατάχ. Θα σας είμαι ευγνώμων εάν μπορείτε να μας πείτε σχετικά κάποιες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ κύριε Λίτς, κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήλθατε κύριε Υπουργέ, κύριε Αλμάλκη. Ε, επιθυμώ να σας πω ότι παρακολουθούμε και από τη χώρα μου πάρα πολύ προσεκτικά το Παλαιστινιακό. Μα απασχολεί πολύ το θέμα τη σύλληψη και κράτηση νεαρών Παλαιστινίων από τις αρχές του Ισραήλ. Έχουμε απευθύνει και έκκληση στον επικεφαλής της αρμόδιας, της αρμόδιας Ισραηλής Καμιά φορά τα παιδιά αυτά κρατιούνται σε διοικητική κράτηση εντελώς ε, εκτός νομιμότητας. Ε, άλλη ερώτηση. Όλες οι διαπραγματεύσεις και συζητήσεις σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους έχουν ανακοπεί. Ποια είναι η γνώμη σας. Ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να ξεπεραστεί αυτή η στασιμότητα. ευχαριστώ. Η κυρία Λιωμαρή, επιθυμώ να ευχαριστήσω για την παρέμβασή του τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης. Όταν ήμουν επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας εδώ και μια πενταετία, είχα επισκεφθεί επισήμως το Ισραήλ και τη Ραμαλά βεβαίως και αυτό που με είχε εντυπωσιάσει τότε στις συζητήσεις μου και με τους πολιτικούς ηθήνοντες αλλά και με τον κόσμο έξω όταν μετακινούμε. Ήταν μια κάποια αντίθεση που υπήρχε ανάμεσα σε έναν κόσμο, ένα κοινό που ονειρευόταν την ειρήνη και την εποχή όπου μπορούσε κανείς να διαβαίνει από τη μια μεριά στην άλλη και η Παλαιστίνη προς τη μεριά του Ισραήλ και η Ισραηλοί προς τη μεριά ε, και της Γάζας ε, για να εορτάσουν και διάφορες μουσουλμανικές εορτές υπήρχε κάποια ελπίδα και υπήρχε κάποια ελπίδα και τότε που είχα επισκεφθεί εγώ για να ξαναβρούν αυτή την κατάσταση από την άλλη μεριά από μια αντιπολίτευση που μου έδειχνε μια εσωτερική ένταση και που αποτελούσε μια τροχοπέδη στην εξέβρεση λύσης. Έχω λοιπόν τρεις ερωτήσεις. Μία η οποία τέθηκε ήδη σε ό,τι αφορά την ικανότητα ενότητας των Παλαιστινίων για την προπαρασκευή των διαπραγματεύσεων. Βρίσκεται, θεωρείται πράγματι ότι οι πολιτικοί ευθύνοντες κάθε είδους έχουν μια πραγματική βούληση προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερο, δεύτερο ερώτημα. Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να πείτε τα πάντα βεβαίως επ' αυτού. Αλλά ποια είναι τα περιθώρια διαπραγματεύσεων που έχετε. Τι μπορείτε να μας πείτε ό,τι αφορά τα διαπραγματευτικά σα περιθώρια. Τρίτη ερώτηση που νομίζω ότι δεν μας απασχολεί επαρκώς. Θα ήθελα να γνωρίζω Ποιο είναι ο ρόλος και ενδεχομένω η θέση των Παλαιστινίων που δεν βρίσκονται στο έδαφος της Παλαιστίνη. αλλά που είναι σε όμορα, κοντινά εδάφη. Παίζουν κάποιο ρόλο. Έχουν θέση έχουν κάποιες θέσεις και απέναντι στις κυβερνήσεις των χωρών όπου διαβιούν, για παράδειγμα η Ορδανία, Λίβανος και άλλες χώρες. Και είναι ενιαία η στάση τους αυτή. Και ποια είναι η στάση τους αυτή απέναντι στις διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι ανάγκες τους και ποια είναι επίσης και από την πλευρά τους τα διαπραγματευτικά περιθώρια. Σας ευχαριστώ. Εσείς κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκόμης. Ποτέ δεν άκουσα και διορθώστε με εάν κάνω λάθος δεν έχω ακούσει καμιά φορά να έχει πει το Ισραήλ ότι παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο ρόλο στη διαδικασία ειρήνευσης. Το Ισραήλ ποτέ δεν είπε ανοιχτά, καθαρά, ότι καλωσορίζει οποιονδήποτε ρόλο της Ευρώπης στην ειρηνευτική διαδικασία Ισραήλ-Παλαιστίνης. Ποτέ. Αυτό που λέει πάντοτε το Ισραήλ Λέει, ποτέ μην κάνετε αυτό, διότι αλλιώ θα χάσετε την πιθανότητα να παίξετε κάποιο ρόλο. Αλλά ποτέ δεν σας έχει προσκαλέσει να παίξετε οποιονδήποτε ρόλο. Το Ισραήλ. Το Ισραήλ πάντοτε βάζει βέτο σε οποιονδήποτε ευρωπαϊκό ρόλο Στη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ Παλαιστινίων. Βάζει βέτο. Και τους προκαλώ να πούν όχι στον ισχυρισμό μου αυτό. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι πάντοτε καλωσορίσαμε τον ευρωπαϊκό ρόλο διότι εμείς πιστεύουμε στην σημασία της Ευρώπης και στο να παίξει ένα ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Είπαμε πάντοτε ότι δεν θέλουμε η Ευρώπη να είναι απλώς payer, δηλαδή να πληρώνει μόνο, αλλά και player, δηλαδή να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε αντιληφθεί από την αρχή το γνήσιο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και επιθυμία να συμμετάσχετε, γιατί εμείς είμαστε στο κάτω-κάτω στην αυλή σας, η αυλή της Ευρώπης οτιδήποτε συμβαίνει σε Ισραήλ-Παλαιστίνη φύγει έμεσα ή άμεσα και την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ναι, κατανοούμε, ναι, προωθούμε, ναι, δεχόμαστε, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε τον ευρωπαϊκό ρόλο. Πάντοτε ζητούσαμε να παίξει ρόλο η Ευρώπη, ενώ το Ισραήλ πάντοτε αποθούσε το ενδεχόμενο αυτό, οποιοδήποτε, ρόλο της Ευρώπης. Πάρουμε τώρα την ε, γαλλική πρωτοβουλία ως παράδειγμα. Αμέσως, αμελητή και χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία δισταγμό, είπαμε ναι. Γιατί, για δύο απλούς λόγους. Πρώτο, διότι η γαλλική πρωτοβουλία έρχεται δύο χρόνια μετά την αποτυχία του Τζον Κέρι να επιτύχει αποτέλεσμα στη διαπραγματεύση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίου. Ενώ τον Μάρτιο του 2014. Τίποτα δεν έγινε στην πραγματικότητα. Δύο χρόνια χωρίς καμιά ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών. Δεύτερο, διότι η Γαλλία είχε το θάρρος να βγει μπροστά και να πει ναι θέλουμε να συμμετάσχουμε διότι ως Γαλλία μπορούμε, μάλλον δεν μπορούμε να καθόμαστε άπραγοι και να παρακολουθούμε την επιδείνωση της καταστάσεως η οποία εν τέλει θα επηρεάσει και εμάς. Ω Γαλλία, ω Ευρώπη, ω κόσμο. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θαραλέα στάση. Και γι' αυτό είπαμε στην Γαλλική Πρωτοβουλία και παρά το γεγονό ότι η Γαλλική Πρωτοβουλία δεν υλοποιήθηκε σωστά, παρόλα αυτά, διότι έχει ακόμα κενά τα οποία πρέπει να πληρωθούν, είπαμε όμω, ναι. Και σπρώξαμε κι εμεί και αρχίσαμε μάλιστα και το λόμπι. Ο πρόεδρο μου σηκώθηκε και πήγε στην Ιαπωνία, Νότια Κορέα και άλλε χώρε. για να προωθήσουμε εκεί την γαλλική πρωτοβουλία και οι χώρες αυτές την στήριξαν και είπαν ότι θέλουν και αυτοί να προσκληθούν. Η Ινδονησία είπε ότι θέλει να προσκληθεί. Και άλλες χώρες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαλλική πρωτοβουλία, διότι είναι η μόνη πρωτοβουλία που υπάρχει. Εάν αποτύχει η γαλλική πρωτοβουλία, τι θα συμβεί, πού πάμε, πού κατευθυνόμαστε, σε ένα πολύ επικίνδυνο κόσμο. Είναι λοιπόν σημαντικό να ενισχυθεί η γαλλική πρωτοβουλία, να συνεργαστούμε με τους Γάλλους για να υλοποιηθεί. Μέχρι τώρα οι Ισραηλοί δεν έχουν ανταποκριθεί, μόνο όρους βάζουν. Και ακόμα περιμένουμε βέβαια τους Αμερικανούς. Μιλήσαμε με τους Αμερικανούς, είδαμε τον Τζον Κέρι προ τριών εβδομάδων στο Αμάν και του μιλήσαμε για τη γαλλική πρωτοβουλία. Μας είπε ναι, την ακούσαμε τη γαλλική πρωτοβουλία και την μελετούμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ανάγκη να εμπλέκεται η Ευρώπη. Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι πολύ σημαντική σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Προφανώς τώρα, σε ό,τι αφορά τη γαλλική πρωτοβουλία, πού βρίσκεται. Συναντήσαμε τον Γάλλο Υπουργό των Εξωτερικών ως μέρος της τετραμερούς στο Κάιρο προ δύο εβδομάδων στις 9 ε, του τρέχοντος μηνός συναντήθηκε μαζί μας, τους υπουργούς εξωτερικών δηλαδή Αιγύπτου, Ιορδανίας, Μαρόκου, Παλαιστίνης και το Γενικό Γραμματεία του Αραβικού Συνδέσμου και μας εξήγησε ο Γάλλος υπέξ τα της Γαλλικής Πρωτοβουλίας και εμείς δηλώσαμε ως Άραβες ότι στηρίζουμε τη Γαλλική Πρωτοβουλία και εξακολουθούμε να το πράττουμε. Προ λίγων ημερών δέχτηκα τον ειδικό απεσταλμένο στη Ραμάλα της γαλλικής κυβέρνησης για τον σκοπό αυτό. Συναντήθηκε μαζί μου με τους Ισραηλινούς, με τον Μαχμού Ταμπάς, πήγε μετά Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και αλλού και αναμένουμε τώρα να λάβουμε κάποια αντίδραση από τη γαλλική πλευρά σχετικά με τα, όσα άκουσε από τους διαφόρους συνομιλητές του, Ουάσιγκτον κλπ. Για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ ως κυβέρνηση, ως χώρα και ως Υπουργείο για να στηρίξουμε τη γαλλική πρωτοβουλία, για να συνεργαστούμε με τους Γάλλους για να μπορέσει να υλοποιηθεί η ιδέα τους. Έχει καταστεί σαφές ότι η γαλλική πρωτοβουλία θα πρέπει να περιέχει κάποια βασικά στοιχεία για τα οποία πρέπει να δοθεί αγωνες δηλαδή πρώτα πρώτα πώς θα προστατευτεί, θα διασωθεί η επιλογή, η λύση των δύο κρατών που τώρα κινδυνεύει. Και γνωρίζουμε τι είπε ο Πρωθυπουργό Κάμεραν ότι ε, σβήνει αυτή η λύση, κλείνει η πόρτα αυτής της επιλογής. Να, μια άλλη πρόκληση που σας θέτω. Ρωτήστε τον Εντανιάχου. Δημοσία υποστηρίζει τη λύση αυτή ή ου. Όχι δεν την υποστηρίζει. Αντιθέτως, ό,τι κάνει, ό,τι οι πολιτικές ασκεί αποφασίζει και υλοποιεί, αποσκοπούν στο να δυναμητήσουν τη λύση των δύο κρατών. Και πέραν αυτού, καθίστε και κοιτάξτε τι δηλώσεις έχουν κάνει οι υπουργοί στην ε, ε, κυβέρνηση συνασπισμού και βλέπετε ότι η δημοσία όλοι τοποθετούνται κατά συγγράφουν άρθρα στο New York Times και σε άλλες εφημερίδες κατά τις λύσεις τούτες. Απεργάζονται λύσεις, ε, πράξεις κατά αυτής της ε, λύσης. Και αφού η κυβέρνηση της χώρας ε, έχει κάθε νομιμότητα, πού είναι ο συνομιλητής μας, Πώς είναι δυνατόν ο συνομιλητής να υπονομεύει, να εκφράζεται, να τοποθετείται κατά της λύσης των δύο κρατών. Να ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Επομένως, η γαλλική πρωτοβουλία για μας είναι μια δυνατότητα του να προστατεύσουμε αυτήν την λύση που ακόμα είναι μια υπαρκτή επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν πρόκειται για κάτι το οποίο μόνο Εμένα θα πρέπει να με νοιάζει και εσείς θα πρέπει να μεριμνάτε για αυτή την λύση γιατί είναι η μόνη διέξοδος. Υπάρχει παγκόσμια συνένεση ότι δηλαδή αυτή είναι η λύση του προβλήματος του Μέσα Ανατολικού. Αν αρθεί, αν καταργηθεί, αν εξαφανιστεί αυτή η λύση, τι θα απομείνει. Είναι επομένως η επιτακτική ενέργεια να προστατεύσουμε αυτή την λύση. Άπαξ και υπονομεύεται αυτή η λύση δεν μένει τίποτα. Ένα κράτος, δύο εθνοτήτων, αυτό θέλει το Ισραήλ. Αυτό είναι κράτος όπου πριν ανέβει το Απαρτχάιν. De facto. Κανείς δεν το ζητάει αυτό. Εμείς θέλουμε να συνεπάρξουμε σε δικό μας κράτος πλάι στο Ισραήλ με ειρήνη και ασφάλεια. Αυτό πάνε να πει για μας λύση των δύο κρατών. Άρα προστατεύστε μας ε, προστατεύστε αυτή τη λύση. Είναι και δικός σας αγώνας, όχι μόνο δικός μας. Και τελικά η άλλη πάργουσα επιλογή είναι ένα και μόνο κράτος δύο εθνοτήτων. Όμως έχουμε από τη μία μεριά τη δημοκρατική λύση και από την άλλη μεριά την αντιδημοκρατική όπου όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Και από πλευράς δημογραφικάς σε μια διετία, τριετία, εμείς θα είμαστε η πλειοψηφία σε αυτό το δημοκρατικό κράτος των δύο εθνοτήτων. Άλλη επιλογή, μη δημοκρατικό κράτος που κυριαρχεί το apartheid. Αυτά πρεσβεύει το Ισραήλ να μας έχει εμάς πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Apartheid που δεν υπάρχει ανοχή, ανεκτικότητα και αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε επομένως γιατί να ξεκινήσουμε έναν τέτοιο αγώνα. Να συνεχίσουμε το σημερινό αγώνα για να προστατεύσουμε τη λύση των δύο κρατών. Αυτό τον αγώνα να δώσουμε που για μας είναι επιτακτικής ανάγκης και πάρα πολύ ε, σημαντική υπόθεση και για μας και για τους Ισραηλινούς και για σας. Πολύ σημαντικό. Άλλο θέμα τώρα γιατί εμείς προωθούμε την γαλλική πρωτοβουλία γιατί μιλά για διαπραγματεύσεις ως τρόπο άρσης των προστριβών και των συγκρούσεων. Μιλά για χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να λάβει τέλος η κατοχή που κρατά μία 48 ετία μιλά για κάποιους όρους αναφοράς για τα 67 σύνορα. Μιλά για το endgame, δηλαδή για Παλαιστινιακό κράτος που θα συμβιώνει στο πλάι, στην πλευρά του Ισραηλινού κράτους. Να, αυτά θέλουμε και σε αυτά συμφωνούμε και αυτό που θα την ελοποιήσει η γαλλική λύση, όλα αυτά μας θέτει επί της τραπέζης, άρα θα πρέπει αυτή την πρωτοβουλία να προωθήσουμε, θα πρέπει να εργαστούμε για αυτή την πρωτοβουλία και δεν θα πρέπει να αφήσουμε να καταπέσει αυτή η λύση γιατί δεν υπάρχουν αλλακτικέ ή τέλος πάντων είναι κάτι το πολύ χειρότερο. Στη γωνία περιμένει το Ισλαμικό κράτος, περιμένει την αποτυχία αυτών των διαδημάτων και είναι πάρα πολλοί Ισραηλοί επίσημοι και εμει οι οποίοι συνεργάζονται έμεσα με το Ισλαμικό κράτος ούτως ώστε να αποτύχει η Γαλλική Πρωτοβουλία. Θα πρέπει να δείτε τη σύνδεση των δύο θεμάτων. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει επομένω να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση τώρα όσον αφορά την νεολαία της χώρας. Αυτή που από απελπισία δεν νιώθουν να υπάρχει καμία ελπίδα και αυτοκτονούν πηγαίνοντας στα φυλάκια στα σημεία ελέγχου των Ισραηλινών και αυτοκτονούν. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, από τότε που ξεκίνησε η επίθεση στους Ελληνούς στρατιώτες με ε, μαχαίρια κλπ. έχουν έτσι σκοτωθεί πάνω από 200 Παλαιστινίους. 80% αυτών ήταν νέοι. 12 με 21. 12 με 21 μάλλον. Και το 80% αυτών που έκαναν αυτές τις επιθέσεις που έγιναν σε αυτά τα σημεία ελέγχου του Ισραηλινού στρατού που βρίσκονται όχι το Ισραήλ αλλά εντός Παλαιστινιακού εδάφους. Οπότε ποιο είναι το ερώτημα γιατί οι Ισραηλινοί φαντάροι να βρίσκονται εκεί. Τι κάνουν. Γιατί να έχουν σημεία ελέγχου στην καρδιά της ε, Παλαιστινιακής επικράτειας. Για ποιο λόγο. Τι δουλειά έχουν εκεί. Γιατί ένας Ελληνός πολίτης που ονομάζεται επικιστής περπατάει, κινείται, οδηγά στην καρδιά της Δυτικής Όχθης. Πολύ βασικό ερώτημα τούτο. Οπότε, ναι, ένας χρόνο όταν τα βλέπει αυτά, ε βέβαια, νιώθει απογοήτευση, νιώθει ματέωση, νιώθει απελπισία, νιώθει να μην έχει μέλλον, νιώθει ότι θέλει κάποιον να δώσει τέλος σε αυτό το τον πόνο και λέει ότι θα πάει και θα επιτεθεί σε αυτό το σημείο ελέγχου το οποίο επανδρώνεται με αυτούς τους πάνωπλους φαντάρους και τους επιτίθεται. Ξέρει ότι η ενέργεια αυτή είναι αυτοκτονική, ότι θα πεθάνει και ξέρει ότι θα σκοτωθεί πριν σκοτώσει κανένα άλλο, αλλά δεν έχει εναλλακτικέ. Δεν έχει όμως και πιθανότητες να βγει ζωντανό από αυτή την υπόθεση. 0% είναι πιθανότητε και το κάνει αυτό ένας 12χρονο το συνειδητοποιείται. Θέλει να αυτοκτονησει ενα ένας 12χρονο που δεν ξέρει τίποτα για τη ζωή ακόμα. Και καταλήγει σε τέτοιο συμπέρασμα ότι η ζωή δεν αξίζει υπ' αυτούς τους όρους. Και βάζει τέλος στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Είναι τρομερό αυτό. Φυσικά και είμαι κατά μια τέτοια συμπεριφορά. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το φαινόμενο. Όμως δεν μιλάμε για καθηγητές πανεπιστημίου, μιλάμε για ψυχολόγους. Πασχίζουν να καταλάβουν τι γίνεται. Αλλά πρόκειται περί της πραγματικότητας και νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η κατοχή. Η κατοχή που θα πρέπει να λάβει τέλος. Θα πρέπει το Ισραήλ να θέσει ένα τέρμα και έτσι να ζουν οι Ισραηλοί καλύτερα. Να υπάρχει ευημερία, να υπάρχει επιβίωση και να υπάρχει συμβίωση και συνύπαρξη μεταξύ γειτόνων φίλων. Με ρωτήσανε επίσης πώς βλέπω την κατάσταση, πώς βλέπω το Ισραήλ, ακριβώς. Έχουμε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Πολύ πριν τη συμφωνία του Όσλο, το 1993. Και από τότε συνεργαζόμαστε με το Ισραηλινό κράτος για θέματα ασφάλειας. Υπάρχει πλήρης συνεργασία μέχρι σήμερα. Πάνω από 20 είναι οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει. Και έχουμε τηρήσει τις δεσμεύσεις μας που απορρίνουν από αυτές τις συμφωνίες και από το Ισραήλ τι ζητούμε τίποτα. Απλώς να αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν από το 67 Δυτική Όχθη και η Ιερουσαλήμ αλλά και από τη Λωρίδα της Γάζας. Οπότε να υπογραφή μια ειρηνευτική συμφωνία είμαστε πρόθυμοι να συνεπάρξουμε πλάι-πλάι και να συνεργαστούμε με το Ισραήλ. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Θα το, το αναγνωρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τους αναγνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει και εκείνοι να μας αναγνωρίσουν. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε αποφασισμένοι, θα πρέπει να καταλάβουν ότι θέλουμε ανεξαρτησία, Αλλιώς ε, δεν μιλούμε σε βάση ισότητα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την αναγνώριση του Ισραήλ, ενώ εκείνοι δεν μας αναγνωρίζουν. Και δεν ε, είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την τήρηση των συμπεφωνημένων, ενώ το Ισραήλ δεν σέβεται. Δεν σέβεται, δεν τηρεί τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και γι' αυτό πήγαμε και βρήκαμε τη Μογκερίνη και άλλους. Τους είπαμε το τι ζητούμε, ότι θα πρέπει οι Ισραηλινοί να σεβαστούν τα όσα έχουν προσυπογράψει, τα όσα έχουν συμφωνήσει από το Όσλο μέχρι σήμερα. Εάν δεν προτίθενται να κάνουν βήματα πρόοδου, αν δεν θέλουν διαπραγματεύσει. Ε, τότε ας μιλήσουμε για την εφαρμογή των συμφωνιών. Των συμφωνιών μεταξύ ημών και εκείνων. Αλλά χρειαζόμαστε και κάποιον τρίτο, εσάς. Εσάς ως παρατηρητές, ως επόπτες της ε, υλοποίησης, του σεβασμού, της τήρησης των συμφωνιών μας με τους Έλληνους και να δούμε ποιος τηρεί και ποιος δεν τηρεί τα συμπεφωνημένα. Πάρα πολύ απλό. Εμείς προωθούμε αυτή την πρωτοβουλία και τι λέει ότι αν αποσυρθεί από τα κατεχόμενα το Ισραήλ από τα κατεχόμενα από το 1967 από το Γκολάν της Συρίας ή από την Πασνική επικράτεια ή την Λιβανινέζικη επικράτεια τότε όλοι οι Άραβες όλοι πρόκειται να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους θα γνωρίσουμε το Ισραήλ και πρέπει να αποκαταστήσουμε τις μοναδικές σχέσεις με το κράτος Ισραήλ εμείς οι Παλαιστίνοι και όχι οι Ισραηλινοί. Θέλουμε αυτή η πρωτοβουλία να προωθηθεί παντού και στο Ισραήλ το προωθούμε. Ναι, όντως θέλουμε να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία και οπότε αυτό μπορεί να γίνει. τα κυριλόγια δηλαδή της Γάζας. Και εγώ, επειδή συμμετέχω στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, έχω πάει εκεί ως Υπουργός Εξωτερικών, έχω πάει στα πλαίσια μιας αποστολής αντιπροσωπείας, επικεφαλής ήταν ο Πρωθυπουργός, πήγαμε επομένω εκεί και ναι, διατηρούμε γραφεία, λειτουργούμε εκεί και έχουμε όντως πρόβλημα με την Χαμάς. Το δέχομαι. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη επιληθεί. Το παραδέχομαι γιατί υπάρχουν ε, παρεμβάσεις εξωγενών παραγόντων, όχι δικών μας. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι εάν η Αλφατάχ και ε, αν αυτοί απομείνουν να χειρίζονται τα πράγματα τότε θα έχουμε μόνο από Χαμάς και Αλφατάχ πρόβλημα θα πρέπει να δούμε πως η Χαμάς ε, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα χειριζόμενοι, χειραγωγώντας το Παλαιστινιακό. Άρα θα πρέπει οι εκείνες οι κυβερνήσεις να μην αναμειγνύονται στις δικές μας υποθέσεις. Θα πρέπει να μας αφήσουν εμάς να λύσουμε το πρόβλημά μας που μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και να έχουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Έχουμε ένα σωρό επαφές που γίνονται στην Τόχα και αντικατοπτρίζουν όλα αυτά. Έχουμε δύο γύρους που έγιναν και τώρα μιλούμε για κάποιον τρίτο γύρο που σύντομα θα γίνει, οπότε λέμε ότι αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας και να τα βρούμε, αυτό θα γίνει σαν κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και ο κύριος Αμπάς, ο πρόεδρος μας ήταν ε, ξεκάθαρος. Είπε ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι ε, υπό αυτές τις συνθήκες. Πρώτα πρώτα να υπάρχει κυβέρνηση εθνικής ε, ενότητας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βρεθεί μέρα, ημερομηνία για κάποιες κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές, γιατί θα πρέπει να ανανεωθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των ηγετών μας. Με εκλογές. Αυτό πιστεύουμε. Ο πρόεδρος μας από την αρχή επιμένει ότι θα πρέπει να γίνουν εκλογές δεν φοβάται τη δημοκρατία ούτε τις εκλογές. Πάρα πολύ περίεργο αυτό για τη Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα αποχωρήσει και θα δώσει σε νέο ηγέτη τη θέση του. Πολύ σημαντικό θα πρέπει να τον εθαρρύνουμε, θα πρέπει προ τα εκεί να πάμε. Τέτοιου ηγέτε να έχουμε και να μην του ε, αποδυναμώνουμε όταν του έχουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είδατε τι έγινε την τελευταία δεκαετία που ήταν στο Ισραήλ στην εξουσία Νετανιάχου. Τι έγινε με τον Μαχμούν Ταμπάς που τον ταπεινώνει ενώπιον του λαού του. Μιλώντας για διαπραγματεύσεις εκείνος. Μιλώντας για το τέλος της βίας. Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να τον αποδυναμώσουν. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι διαπραγματεύσεις και τέτοιες διαδικασίες δεν ωφελούν δεν αποδίδουν αποτελέσματα. Ουσιαστικά αυτό αβαντάρει τη Χαμάς και τους εξτρεμιστές, τη βία και την στρατιωτική αντιπαράθεση. Έχω πέντε λεπτά ακόμα για να ολοκληρώσω. Δύο, καλώς. Όταν μιλάμε τώρα για τους επικισμούς, οι επικισμοί. Τι είναι. Η πολιτική αυτή δεν είναι απλώς κατάσχεση γης. Η επικιστική αυτή πολιτική δεν είναι απλώς οικοδόμηση επικισμών και μονάδες οικιστικές για τους επίκους. Η επικιστική αυτή πολιτική είναι συλλογική, δηλαδή γίνεται κατάσχεση από γη δηλαδή παίρνουν από ανθρώπους που τους διώχνουν από τα σπίτια τους και βάζουν επίκους στη θέση τους. Είναι μια παραβίαση της σύμβασης της Γενέβης αυτή. Συνεπώς, όταν μιλάμε για επικισμούς, πρέπει να το δούμε σαν μια ολόκληρη επιχείρηση. Κάποιος ο οποίος την φτιάχνει, την προστατεύει, την νομιμοποιεί, κάποιος ο οποίος ε, φτιάχνει και νόμους για να την προστατεύσει αυτή την επιχείρηση, την επικιστική. Αν λοιπόν οι επικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τότε και οι έπικοι είναι παράνομοι. Τότε τα προϊόντα από αυτές τις περιοχές ε, όπου ζουν οι επικισμοί είναι παράνομα. Οι εξαγωγές τους, ό,τι βγαίνει από εκεί δηλαδή, από αυτές τις περιοχές. Και εδώ μιλάμε για τις σήμε των προϊόντων αυτών, για τις ετικέτες που θα τους βάλουμε, όχι απλώς να τα απαγορεύσουμε, αλλά να τους βάλουμε και ετικέτες ώστε, αν μη τι άλλο, να ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το δούμε αυτό και να καταλάβει ο κόσμος, να αντιληφθεί τι αγοράζει τελικά και τι καταναλώνει. Γιατί πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ναι. Είχαμε ανοιχτά σύνορα, Είχαμε μετακινήσεις Ισραηλινών Παλαιστινίων πριν από πολλά χρόνια. Και ήταν προπτικές τότε, πραγματικές για να βρεθεί κάποια λύση. Όταν όμως έγινε περιορισμός στη μετακίνηση των ε, Παλαιστινίων, 600 φυλάκια ελέγχου, και όταν μας ανάγκασαν να έχουμε άδειες να, τέτοιες άδειε. Για να μπορούμε να μετακινούμεθα οπουδήποτε. Άδεια από τις αρτητικές αρχές του Ισραήλ για να μπορούμε να μετακινούμεστε από το ένα σημείο στο άλλο. Χωρίς αυτό το χαρτί δεν μπορούμε. Να, εδώ είναι η φωτογραφία μου, το όνομά μου και λέει ακριβώς τι ώρα, πότε μπορώ να μετακινηθώ από το ένα σημείο στο άλλο. Πώς σας φαίνεται αυτό. Αυτό όμως που λέμε να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση, ναι, όταν μπορούμε να συνεπάρχουμε με τους Ισραηλινούς. Αλλά αυτό γίνεται μόνο αν υπάρχουν οι ίσοι όροι, όταν είμαστε κι εμείς ελεύθεροι όπως είναι και αυτοί, όταν έχουμε την ελευθερία να μετακινούμεθα όπως έχουν και αυτοί. Όχι αν υπάρχουν δρόμοι για αυτούς και άλλοι δρόμοι για μας, αποκλειστικοί δρόμοι για τους Ισραηλινούς και άλλοι που είναι αποκλειστικά για τους Παλαιστινίους, Άλλε άδειε για του μεν, άλλε για του δε, άλλα περάσματα για του μεν και άλλα για του δε. Αυτό μου θυμίζει την Νότια Αφρική πριν από μερικά χρόνια. Εμεί δεν θέλουμε να πάμε πίσω σε αυτή την κατάσταση apartheid. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για όλου, για του ίδιου του Ισραηλινού. Αν θέλουν να σταματήσει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να σταματήσει η κατοχή τους και ό,τι φέρνει η κατοχή αυτή μαζί. Μίσος και περισσότερο μίσος, αίμα και περισσότερο αίμα. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Αν κάποιος φταίει, φταίει η κατοχή. Εγώ δεν τα βάζω με έναν άνθρωπο ή με έναν άλλον, τα βάζω όμως με την κατοχή ως σύστημα. Γιατί αυτό το σύστημα της κατοχής είναι που μας καταστρέφει. Και όταν λέω μας, ενώ εμάς τους Παλαιστινίους, αλλά και εμάς τους Ρελινούς. Όλους μας καταστρέφει η κατοχή. Και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον και να γλιτώσουμε από αυτή την κατοχή που υπονομεύει την ειρήνη και την συνύπαρξή μας στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Αυτή την ε, τόσο ιδιαίτερη μέρα σας ευχαριστώ που ήρθατε και ακούσαμε τις απόψεις σας όσον ε, αφορά τη Γαλλική Πρωτοβουλία και τις προσπάθειες που γίνονται από τη συμφωνία του Όσλο προκειμένου να βρεθεί λύση. Ε, κύριε Μπορκέζιο, θέλατε να πάρετε το λόγο, αλλά ήρθατε αργότερα. Τώρα τελειώνουμε, βλέπετε. Η συνεδρίαση τελειώνει. Μα έδωσε την απάντηση ο Υπουργό. Μισό λεφτάκι μου, μισό λεφτάκι. Ε, να χαιρετήσω τον κύριο Υπουργό και θα πρέπει να καταδικάσουμε το γεγονός το ότι ήρθε εδώ να μας πει για την Ιντιφάντα των μαχαιριών και νομίζω ότι υπό τις σημερινές συνθήκες θα έπρεπε να έχει περισσότερο σεβασμό για αυτό το Πάσχα το Πάσχα που χρησιμοποιείται από την αιματοχυσία που επέβαλαν ε, αυτή οι σφαγείς εδώ στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ευχαριστώ τον Υπουργό. Η επόμενη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ θα λάβει χώρα στις 4 Απριλίου. Σήμερα το απόγευμα δεν υπάρχει συνεδρίαση όπως είπε νωρίτερα και ο Πρόεδρος.